Καλημέρα κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν, ε, να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ακρόαση και θα μιλήσω γερμανικά. Σας καλωσορίζω όλους. Σήμερα ξεκινάει η δημόσια εργασία της Επιτροπής ε, Παναμά στις 14 Σεπτεμβρίου αποστήλαμε την πρόσκληση στους συναδέλφους. Υποθέτω ότι δεν είχαν συντηρήσεις με την ε, διαδικασία διεξαγωγής που προτείνουμε, δεν βλέπω. Οπότε να κάνω μερικές βασικές παρατηρήσεις. Πρώτον, συνολικά έχουμε 18 γλώσσες, άρα όλοι μπορείτε να μιλήσετε την ε, μητρική σας γλώσσα, αν και τα έγγραφα υπάρχουν στα αγγλικά βεβαίως. Δεύτερον, έχουμε έγγραφα τα οποία αποστήλαμε στους συναδέλφους, ε, οπότε δεν θα τα ξαναδιανύμουμε, πρέπει να τα έχετε μαζί σας. Τρίτον, η συνεδρίαση σήμερα μεταδίδεται ζωντανά μέσω του διαδικτύου, υπάρχει web streaming δηλαδή, έχετε τη διεύθυνση του ιστοχώρου και οποιοδήποτε μιλάει, ο κάθε μιλητής ε, θα ε, κινηματογραφείται. Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι συντονιστές έχουν κάποια επιθυμία. Όχι. Ωραία. Α, ο κύριος Ροσάτη συντονιστής του ΕΛΚΑ. Ναι θέλω να πω τυπικά ότι δεν έχουμε συμφωνήσει για τη σειρά των ομιλητών για την ε, συνεδρίασή μας από ό,τι κατάλαβα είναι υποσυζήτηση και θέλω να πω ότι θεωρώ ότι η διαδικασία που εφαρμόζουμε σήμερα είναι κατεξαίρεση μέχρι να καταλήξουμε στην τελική σειρά των ομιλητών από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ κύριε Ροζάτη, λέει ο Πρόεδρος. Το σημειώνω, αλλά πρέπει να υπάρχει κατανόηση. Ο Πρόεδρος έπρεπε να είναι αντικειμενικός, αλλά υπάρχουν κάποιες ασάφειες στο κατάλογο των ομιλητών και είπαμε ότι μετά την πρώτη ακρόαση θα ξανασυζητήσουμε τη σειρά, χωρίς να κάνουμε μια συζήτηση εκβάθρων. Παρακαλώ, ποιο άλλο ζήτησε το λόγο για τη διαδικασία. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την ημερήσια διάταξη. Δυστυχώς, λόγω των αεροπορικών καθυστερήσεων, δεν μπόρεσα να πω στη στη γραμματεία το αίτημα για να λάβω το λόγο. Θα μπορούσατε λοιπόν, ε, αν μπορείτε να το καταγράψετε, θέλω και εγώ το λόγο στη συζήτηση. Αν σας κατάλαβα, δεν λάβατε τα έγγραφα, είπατε. Α, όχι. Τι είπατε. Α. Δυστυχώς το μικρόφωνο του Προέδρου δεν ακούγεται. Τώρα ακούγεται. Ωραία. Να περάσουμε τώρα στην παρουσίαση του θέματος. Καλωσορίζω τους ε, συναδέλφους δημοσιογράφους ε, που είναι παρόντες. Χαιρόμεθα ιδιαίτερα που έχουμε τη δυνατότητα στην πρώτη συνεδρίασή μας να συζητήσουμε για το υπόβαθρο των εγγράφων του Παναμά. Εν τω μεταξύ, ε, ακούσαμε και άλλα στοιχεία από τις Μπαχάμες που και αυτά θα πρέπει να μας απασχολήσουν επειδή είμαι πολλά χρόνια ευρωβουλευτής θυμάμαι την ακρόαση της κυρίας Νέλη Κρούζ το 2004 για να επιβεβαιωθεί ως Επίτροπος για την Ανταγωνιστικότητα και τότε μας παρουσίασε 37 οργανισμούς στους οποίους είχε εργαστεί την ε, προηγούμενη δεκαετία. Μας είχε διευκρινίσει ότι δεν έχει πια καμία θέση σε αυτούς τους φορείς. Και αυτό σημαίνει, με τα στοιχεία που βλέπω τώρα, ότι δεν μας είπε την αλήθεια. Θα πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό. Και υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που το θυμούνται και μπορούν να επιβεβαιώσουν αυτό που είπε. Αν το ξέραμε αυτό που ξέρουμε τώρα, τότε δεν θα είχε πάρει την πλειοψηφία 24-23 που της επέτρεψε να επιβεβαιωθεί ως Επίτροπος Ανταγωνισμού. Πρώτα απ' όλα όμω, θέλω να καλωσορίσω λοιπόν τους δημοσιογράφους. Έχουμε τον Φρέντριχ Όμπερ Μάια από την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung ο οποίος ε, είναι σε επαφή μαζί μα με την Skype, ο Κριστόφ Κλέριξ από το περιοδικό ΚΝΑΚ του Βελγίου, Όλιβερ Τσίλμαν από την εφημερίδα Le Matin Dimanche της Ελβετίας, Γιούλια Στάιν και Γιάνν Στρότσικ από τη Γερμανία, από τη βορειογερμανική ραδιοφωνία, και τη Μίνα ε, Κνούς από την Φινλανδική ε, ραδιοτηλεοπτική οργάνωση. Τους καλωσορίζω όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εργασία σας και για την παρουσία σας. Για μας ε, είναι πολύ σημαντική η εργασία αυτή που κάνετε και ιδιαίτερα για θέματα φορολογίας είναι σημαντικό να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος. Έχουμε λοιπόν ε, ήδη κάνει μέσω των Επιτροπών τάξη 1 και 2 ε, έρευνες για αυτά τα θέματα σε επίπεδο κρατών και μεγάλων οργανισμών, αλλά πρέπει να ερευνήσουμε και σε επίπεδο φυσικών προσώπων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η εργασία σας. Θέλουμε μέσω της ακρόασης σήμερα να καταλάβουμε πώς ε, η ένωσή σας που έχει έδρα στη Washington, η ένωση των δημοσιογράφων που διεξάγουν έρευνες, πώς εργάζεται, σε τι βάση εργάζεται, θέλουμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από τα έγγραφα του Παναμά, θέλουμε να μάθουμε τι δυνατότητες νομοθετημάτων θα μας παρουσιάσετε και τι ρόλο, και τι ρόλο μπορούν να παίξουν διάφοροι που μπορούν να διερευνήσουν ή παίζουν ρόλο γενικότερα. Δηλαδή οι τράπεζες ή δικηγόροι και ιδιαίτερα αυτή η εταιρεία δικηγόρων Mossack Fonseca. Και θα ήθελα να μας πείτε και τι προσδοκίες έχετε έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι συνομοθέτης της Ένωσης. Η αποστολή μας, η οποία εγκρίθηκε από την ε, Ολομέλεια τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Η εντολή μας λοιπόν είναι με τι τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη, όχι συγγνώμη, να διερευνήσουμε σε τι βαθμό κάποιοι φορείς τα κράτη-μέλη δεν τήρησαν ε, τον νόμο και επίσης θέλουμε να μάθουμε εάν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις όλων για να καταπολεμάται η φοροδιαφυγή και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ούτως ώστε να επιτύχουμε αποτελέσματα στην εργασία αυτή. Μία σύντομη τώρα τοποθέτηση για την γνωμοδότηση που απέστειλε η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο με βάση τις ε, διατάξεις για την διεξαγωγή των εργασιών των ερευνητικών επιτροπών και επειδή τα κείμενα αυτά έχουν ήδη, τα κείμενα που έχουμε για τα θέματα αυτά είναι ήδη αρκετά παλιά και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και δημοσίευση των σχετικών εγγράφων. Δεν το έχουμε επιτύχει ε, πλήρως. Είμαστε συζητήσεις με τον, τους επιτρόπους ε, Μοσκοβισή και Γιούροβα και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν ε, νέοι κανόνες. Γιατί η έκθεση Κορμπέτ για τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών των ερευνητικών επιτροπών έχει παγώσει. Ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ελέγχει τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί όπως ξέρετε μπορούμε και να απολύσουμε την Κομισιόν, όπως έγινε κάποια στιγμή. Και γι' αυτό θέλουμε να αναπτυχθεί περισσότερο το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να διεξάγει ε, Τέτοιε εργασίε ερευνητικών επιτροπών και με αυτό συμφωνούν και πολλά εθνικά κοινοβούλια. Βεβαίω ο χρόνο πιέζει, αλλά να πω ακόμη ότι έγιναν δύο συνεδριάσεις των συντονιστών για να προετοιμάσουμε την εργασία εδώ και επίσης παραγγείλαμε και ορισμένες ε, μελέτες και θα λάβουμε υπόψη και όλες τις μελέτες που έχουν κάνει οι επιτροπές τάξη 1 και 2 και έχουμε προγραμματίσει μια σειρά ακροάσεων λοιπόν και επισκέψεις ε, σε διάφορα κράτη-μέλη. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν τελειωτικά ακόμη αποφασιστεί η Επιτροπή μας. Πάνα λοιπόν είναι υποχρεωμένη να εργαστεί με τρόπο διαφανή και οπωσδήποτε θα γίνει αυτό. Έχουμε και ένα ειδικό ιστοχώρο όπου θα δημοσιευθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες, όλες οι ακροάσεις και συνεδριάσεις Επιτροπής επίσης θα είναι δημόσιες, ούτως ώστε όλοι να μπορούν να τα παρακολουθήσουν. Τέλος. Όπως συμφωνήσαμε, ακούσατε ήδη την ε, παρέμβαση του συναδέλφου Ροσάτη. Σήμερα λοιπόν έχουμε πέντε ομιλητές στις Βρυξέλλες. Ένας ομιλητής θα μας μιλήσει μέσω βίντεο διάσκεψης. Θα ξεκινήσουμε με δύο εγγεγραμμένα μηνύματα, δύο βίντεο, δύο δημοσιογράφων που δεν μπορούν να παρευρεθούν σήμερα. Είναι μαγνητοσκοπημένα μηνύματα. Κάθε ομιλητής έχει 7 λεπτά για την παρουσίασή του. Μετά την παρουσίαση των ομιλιών, μετά όλες τις ομιλίες, θα υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής μας Οι ερωτήσεις θα γίνονται ανά πεντάλεπτον και ο κάθε ομιλητής θα έχει ένα λεπτό στα πλαίσια αυτού του πενταλέπτου, μετά θα υπάρχουν απαντήσεις και αν επιτρέπει ο χρόνος θα υπάρχουν και περαιτέρω ερωτήσεις. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι και ε, ακριβείς και στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις ούτως ώστε να μην χρειαστεί να σας διακόψει ο Πρόεδρος. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα με τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα του Gerald Βάιλ και της Μαρίνα Δόκαλ. Ο Gerald Βάιλ που είναι επικεφαλής του Διεθνούς ε, Ομίλου των ερευνητών δημοσιογράφων που έχει ε, την έδρα της στην ε, Washington DC. Και επίσης μετά θα ακούμε τον κύριο Obermeier που είναι της Süddeutsche Zeitung και είναι επίσης στην Washington γιατί τώρα πλέον μετά τη δημοσίευση των εγγράφων του Παναμά είναι τη της Deutsche στην Washington. Ξεκινάμε λοιπόν με την ε, βίντεο διάσκεψη. Όπως βλέπετε είναι όλα έτοιμα. Παρακαλώ. Washington, D.C. Yeah. And what we do is we bring investigative... Είμαι ο Τζέραλτ Ράιντ, διευθυντή του Διεθνού Κονσόρτσιουμ των Ερευνητών Δημοσιογράφων. Το Ίδρυμά μα είναι μη κερδοσκοπικό οργανισμό με βάση το Washington DC. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι φέρνουμε μαζί του ερευνητέ δημοσιογράφου για να εργαστούμε σε θέματα τα οποία ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα. Και συνεργαζόμαστε για τα ζητήματα αυτά. Έχει πέρασει ένα χρόνο από τότε που η Deutsche Zeitung ο εταίρος μας στη Γερμανία, μας έφερε 11,5 εκατομμύρια έγγραφα που είχαν πάρει από κάποιον ανώνυμο, ε, κάποιο ανώνυμο άτομο. Τα έγγραφα αυτά ήταν τα αρχεία 40 ετών της Παναμαϊκής νομική, ε, Εταιρείας Νομικών Συμβούλων Μοσάκ Φονσέκα. Εμείς δώσαμε τη δυνατότητα σε 76 οργανισμούς μέσω ενημέρωσης από σε οργανισμούς από 76 χώρες να εργαστούν για αυτά τα έγγραφα και να δουν υπάρχει κάποιο δημόσιο ενδιαφέρον για αυτά τα έγγραφα. Αυτό που βρήκαμε ήταν σοκαριστικό. Πάνω από 140 εκλεγμένοι αξιωματούχοι είχαν εταιρείε υπεράκτιε. Δεν ήταν όλα αυτά τα οποία βρήκαμε παράνομα ή αθέμητα, αλλά <clears throat> αυτό που βρήκαμε ήταν ο μεγαλύτερος όγκος εγγράφων που παρέχουν εσωτερικές πληροφορίες για το σύστημα των φορολογικών παραδείσων. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν τώρα είναι ότι η κοινωνία των πολιτών έχει αντιδράσει στα ευρήματά μας και η ακρόαση αυτή σε κοινοβουλευτικό επίπεδο είναι ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία χαιρετίζουμε. Πρέπει ως δημοσιογράφοι να αποκαλύπτουμε όλα αυτά τα οποία είναι λάθος στην κοινωνία μα και η κοινωνία των πολιτών και οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι θα πρέπει να κάνουν όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα στη συνέχεια και γι' αυτό σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ράιλ. Περνάμε στο μήνυμα του κυρίου Ομπερμάιερ.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 είναι μεγάλη μου ε, χαρά όταν έλαβα το πρώτο μήνυμα από τον πληροφοριοδότη τη υπόθεση Panama Papers. Το πρώτο του μήνυμα ήταν σαφέ. Είμαι ο κύριο Τάδε, που σε ενδιαφέρουν τα στοιχεία που έχω. Όταν το διάβαζα το μήνυμα αυτό, μια χειμωνιάτικη νύχτα πριν από ένα χρόνο, ε, θεώρησα ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί μιλάει για μυστικά στοιχεία εταιριών offshore και με πολλά δεδομένα. Ήταν πολύ παραπάνω από αυτό όμω. Στην πραγματικότητα, άλλαξε και τη δική μου τη ζωή και τη ζωή του συναδέλφου μου, του Φρέντερικ Όμπερμαγερ. Λίγους μήνες μετά εργαζόμασταν από την οργάνωσή μας και με εκατοντάδες από τους καλύτερους ερευνητές δημοσιογράφους παγκοσμίου στη μεγαλύτερη ε, ομάδα συνεργασία ε, δημοσιογράφων ε, που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Μια τεράστια προσπάθεια για να συγκεντρώσουμε δεδομένα, αλλά και τη μεγαλύτερη διαρροή που είχαμε δύο τώρα στον, στη δημοσιογραφία. 2,6 τεραμπάιτ εσωτερικών, εσωτερικών αδελαχθέντων email εγγράφων, ε, συμβάσεων, τραπεζικών δεδομένων και ακόμη και αντιγράφων διαβατηρίων. Έδειχνε πως πολιτικοί, εγκληματίες και πάρα πολλοί φοροφυγάδες κατάφεραν να κρύψουν τα ίχνη τους και μεγάλες τράπεζες ε, τους βοηθούσαν με μεγάλη χαρά. Βρήκαμε στοιχεία για 70 τουλάχιστον πρώην αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Κάποιε κυβερνήσει πραγματικά κλονίστηκαν και υπήρξαν μαζικέ διαμαρτυρίε σε διαφορετικέ χώρε με την παρέτηση του Πρωθυπουργού τη Ισλανδία ω πρώτο δείγμα, αλλά και πολλού υπουργού και τραπεζίτε καθώ και πολλέ έρευνε παγκοσμίω. Ελπίζουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα μπορέσει να φωτίσει ακόμη περισσότερο αυτή την υπόθεση στον κόσμο και θα ε, ρίξει φως ακριβώς αυτήν την παράλληλη πραγματικότητα όπου οι υπερβολικά πλούσιοι και ισχυροί μπορούν να αποφεύγουν τους ε, φόρους και τους νόμους. Αυτό είναι πραγματικά άδικο και πρέπει να σταματήσει. Οι κανόνε που έχουμε συμφωνήσει πρέπει να ισχύουν για όλου. Και για του υπερβολικά πλούσιου, που είναι το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού, και για του υπόλοιπου, που είναι το 99%. Ιδάλω, η δημοκρατία κινδυνεύει οι λαοί και οι άνθρωποι θα χάσουν την πίστη του στη δημοκρατία και δεν ξέρουμε τι θα γίνει εάν η δημοκρατία πραγματικά χαθεί. Οι άνθρωποι ψηφίζουν και να έχουν απλέ λύσει, αλλά τελικά ψηφίζουν και για λαϊκιστέ, για ρατσιστέ και για φασίστε. Σα εύχομαι καλή τύχη λοιπόν και επιμονή για την έρευνα αυτή το διεθνέ λόμπι της ε, χρηματοοικονομία δεν θα σας συμπαθήσει, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε όχι μόνο για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ και τις ευχέ μου για καλή τύχη από τον Ανάρμπο στο Μίσιγκαν. Äh, σας ευχαριστώ. Έχουμε δει λοιπόν τα σχόλια των δύο αυτών δημοσιογράφων. Χαιρόμαστε για τη δυνατότητα που είχαμε να ακούσουμε, έστω και έμεσα, τις απόψεις τους και μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε με τους ομιλητές που προβλέπονται στο πρόγραμμα. Πέντε ομιλητές. Ο πρώτος είναι συνδεμένος μέχρι του Skype, ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσουν καλά και λογικά θα είναι σε θέση να απαντήσει και στα ερωτήματά σας. Θα παρακολουθήσει το σύνολο της συνεδρίασης από το Skype ο Φρέντε Κόμπερμαρ, αλλά με αι, όχι α, όπω όπως ο προηγούμενος ομιλητής, για να υπάρχει και η διαφορά. Λοιπόν, δεν πρέπει να τους <laughs> μπερδέψετε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την ε, βιντεοδιάσκεψη με τον κύριο Ομπερμάιερ με «Η». Dear Mr. Lamming, dear Ελπίζω ότι θα μπορέσω να συμβάλλω σε κάποιο βαθμό στην ε, ε, συνάντηση αυτή. Μήπως μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά, λέει ο πρόεδρος, κύριε Ομπερμάιερ. Πρόκειται για εγκληματίες οι οποίοι συγκαλύπτουν αυτά τα οποία κάνουν μέσω εταιριών offshore ο εξάδελφος του Μπασάρ Αλασάντ, παραδείγματος χάρη, μπορεί να ξεπεράσει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν τον τρόπο. Και αναφερόμαστε στα έγγραφα του Παναμά γιατί η εταιρεία Mossack Fonseca που είναι στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας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 απεσυνδέθη ο κύριος Ομπερμάιερ, αλλά ελπίζω ότι μπορεί να μας ακούσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ομπερμάιρ. Μας ακούτε? Βλέπουμε μία ακίνητη εικόνα από τη δική σας πλευρά. Ίσως θα προσπαθήσουμε και αργότερα να επανακαστήσουμε την επαφή. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κανονικά, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά κανονικά λειτουργεί πολύ καλύτερα το σύστημα. Σας παρακαλώ, όπως έχουμε συμφωνήσει, να παραμείνετε συνδεδεμένος και ε, ή δυνατόν απαντήσετε στις ερωτήσεις. Συνεχίζουμε τώρα. Και έρχομαι στον επόμενο ομιλητή, Κρίστοφ, Κρίστοφ Κλέριξ από το Βέλιο, από το ΚΝΑΚ. Ο κύριος Κλέριξ θα έχει 7 λεπτά στη διάθεσή του. Παρακαλώ κύριε Κλέριξ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω για 7 λεπτά για την έρευνα που έχουμε κάνει στο Βέλιο. Ήταν συνεργασία μεταξύ του Details, Knack και Soir. Όπως ελέγχθη πρόκειται για κάπου 11,5 εκατομμύρια έγγραφα, κάποια από τα οποία έχουν να κάνουν με το Βέλιο και υπάρχουν 732 πολίτες ή κάτοικοι του Βελίου οι οποίοι εμπλέκονται οι οποίοι συνδέονται σε πάνω από χίλιε εταιρείε offshore. Λέω πολίτε του Βελγίου, 1.144 εταιρείε, γιατί υπάρχουν διαφορετικέ εθνικότητε. Έχουμε και Γάλλου και Ολλανδού και από άλλε χώρε. Ε, τα βρετανικά νησιά της Παρθένου είναι ο κύριος προορισμός του ως φορολογική παράδειση, αλλά και ο Παναμάς, και εδώ βλέπετε το έγγραφο αυτό στα Virgin Islands, στα βρετανικά Virgin Islands, όπου υπήρχε και το γραφείο της Μοσάκ ε, Φονσέκα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους Βέλγους, τους υπεράκτους Βέλγους όπως λέμε ζούσαν στην Αμβέρσα και στις Βρυξέλλες. Και ήταν μέτοχοι, ήταν εξουσιοδοτημένοι διευθυντές και είναι περίπου 80, είναι περίπου 80 αυτοί οι οποίοι είναι τελικοί δικαιούχοι. Αυτό το οποίο συμβαίνει με τις εταιρείες οι οποίες είναι offshore είναι ότι δημιουργούνται σε μια χώρα που έχει χαμηλό φορολογικό επίπεδο, αλλά το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να καταλάβετε είναι ότι οι εταιρείε offshore οδηγούν στην ανοημία. Μπορείτε να φτιάξετε μια εταιρεία και να μείνετε εσεί ανώνυμο ω πραγματικό δικαιούχο. Έχουμε 80 λοιπόν τελικού δικαιούχου και αυτό σημαίνει την σημασία αυτού του εγγράφου το οποίο ήρθε στα χέρια μα. Των εγγράφων καλύτερα γιατί αυτοί είναι οι τελικοί δικαιούχοι, αυτοί οι οποίοι παραμένουν άγνωστοι και ανώνυμοι, διότι καλύπτονται πίσω από ε, εμφανιζόμενους ως μετόχους και διευθυντές. Κάποιες λοιπόν από τις περιπτώσεις που ανακαλύψαμε έχουν να κάνουν με τις πιο πλούσιες οικογένειες στο Βέλιο και έχουν ήδη εμφανιστεί σε άλλες έρευνες όπως το LuxLeaks και το SwissLeaks. Επί τη βάση της ανάλυσης των δεδομένων μπορούμε να βρούμε και ποιο ήταν το προφίλ αυτών των Βέλγων πολιτών οι οποίες είχαν μια τέτοια υπεράκτια εταιρεία και φυσικά πολλοί από αυτούς ήταν από το χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά δεύτερη σε σειρά ερχόταν η, ο κλάδος επεξεργασίας διαμαντιών και αυτό το έχουμε αναφέρει σε διάφορα άρθρα για μια ακόμα φορά ο τομέας αυτός των διαμαντιών ήταν ένας τομέας ο οποίος ήταν πολύ προεξάρχον και μέσα στις έρευνες των Links. Υπήρχαν λοιπόν 65 διαμαντάδες οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις ε, υποθέσεις offshore. Έχουν δημιουργήσει αυτές τις εταιρείες με δεκαετία του 2000 με κορύφωση στο 2004 και αν δείτε πώς ήρθαν σε επαφή με την ε, Mossack Fonseca αυτό έγινε μέσω ελβετικών εταιριών. Υπήρξαν διάφοροι ενδιάμεσοι, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο για να βοηθήσουν του Βέλγου αυτού πολίτε να δημιουργήσουν τι εταιρείε offshore και έχουμε δύο μονοπάτια ουσιαστικά, ένα μέσω Ελβετία και ένα μέσω ε, Λουξεμβούργου. Μια άλλη περίπτωση για την οποία αναφερθήκαμε στο Βέλγιο είναι η προηγούμενη μια εταιρεία που ήταν θηγατρική της Δέξια. Ξέρετε ότι η Δέξια ήταν μια μεγάλη, ένας μεγάλος τραπεζικός όμιλος στο Βέλγιο και είχαν μια θηγατρική στο Λουξεμβούργο που ήταν BAF Λουξανβού και είχε μία άλλη αυτή τη γατρική που λεγόταν Experta Corporate and Trust Services, μια εταιρεία στο Λουξεμβούργο, η οποία έπαιξε το ρόλο του ενδιάμεσου μεταξύ του τελικού πελάτη και της Mossack Fonseca. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον τώρα είναι ότι η εξπέρτα στην ανάλυση που κάναμε ως ε, ερευνητές δημοσιογράφοι ήταν η πρώτη εταιρεία η οποία δημιούργησε υπεράκτιε εταιρείε. Πάνω από 1.600 εταιρείε έχουν δημιουργηθεί από την Εξπέρτα τα τελευταία χρόνια. Και την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύσαμε τα έγγραφα που διέρευσαν από τις Μπαχάμες στο ΚΝΑΚ και εκεί πάλι είδαμε να υπάρχουν ε, εταιρείε οι οποίες δημιουργήθηκαν μέσω της ε, Ελβετικής Οδού στις Μπαχάμες. Επομένως και εκεί η εξπέρτα έπαιξε κάποιο ρόλο στο, στις αποκαλύψεις για τις Μπαχάμες. Και σας υπενθυμίζω ότι ήταν τμήμα του ομίλου Δέξια μέσω αυτής της τράπεζας του Λουξεμβουργού. Και ξέρετε ότι ο, όμιλο όμιλος Δέξια έχει διασωθεί με λεφτά φορολογουμένων στο Βέλγιο. Και είναι ενδιαφέρον ακριβώς να καταλάβει κανείς ότι αυτός ο τραπεζικός όμιλος έπαιξε ένα τόσο μεγάλο ρόλο στη δημιουργία εταιριών offshore σε φορολογικούς παραδείσους. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα έγγραφα τα οποία καταδεικνύουν ότι υπήρξε εμπλοκή τη Εξπέκτα. <clears throat> Ένα από τα έγγραφα αυτά ήταν η λεγόμενη έκθεση επαφή που ε, συντάχθηκε από την Μόσακ Φονσέκα και από το κεντρικό γραφείο της Εξπέκτα στο Βέλγιο. Βλέπετε εδώ ένα email που λέει ότι η Εξπέρτα δίνει όλες αυτές τις υπηρεσίες επί τη βάση του ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου. Είναι η απάντηση που παίρνουμε, η στάνταρ απάντηση που παίρνουμε όταν έχουμε να έρθουμε σε επαφέ και να ερευνήσουμε εταιρείε οι οποίε εμπλέκονται σε τέτοιε υποθέσει. Δεν πρόκειται λοιπόν μονάχα για, τον, για την ΔΕΞΗ, αλλά και η προηγούμενη. Ο όμιλο τραπεζών Φόρτη εμπλέκεται στη δημιουργία <clears throat> τέτοιων εταιριών Μία από αυτές ήταν η Fortis Intertrust. Όταν ήρθαμε σε επαφή με αυτούς, είδαμε κάποια παραδείγματα, τους δώσαμε μερικά από τα παραδείγματα που είδαμε στα δεδομένα και είπανε ότι όταν ήταν μέσα στη διοίκηση της Fortis καλύπταν τις ανάγκες μερικών χιλιάδων εταιριών offshore. Αυτό σημαίνει ότι τα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα της Μόσακ Φονσέκα είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι εμπλέκονται στη δημιουργία εταιριών offshore. Ο αντίκτυπος τώρα των πάνω από 20 άρθρων που δημοσιεύσαμε στο, στο Βέλγιο και σε, άλλα, σε άλλες χώρες, καταρχήν έχουν ξεκινήσει από τις φορολογικές αρχές έρευνας, από τους 732 που εμπλέκονται στον κατάλογο μας, 239 έχουν τύχει ε, έρευνας για από τις φορολογικές αρχές του Βελγίου. Δεύτερον, μια δεύτερη συνέπεια είναι ότι και το Βελικό Κοινοβούλιο ξεκίνησε μια επιτροπή έρευνας για τα έγγραφα του Παναμά και επίσης έχει ξεκινήσει η Βελική Κυβέρνηση διαπραγματεύσει με τον Παναμά για να μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών και τέλος <clears throat> σε ό,τι αφορά τα, τον αντίκτυπο, η εισαγγελική αρχή των Βρυξελών έχει ξεκινήσει μια δικαστική έρευνα στα θέματα αυτά. Δυστυχώς δεν μπορούν να μας δώσουν περισσότερα ε, στοιχεία, διότι είναι εν αυτή η δικαστική έρευνα. Θα ήθελα να κλείσω με το να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή τύχη και να τονίσω την ανάγκη να υπάρχει προστασία των καταγγελόντων, των whistleblowers. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μιλούσαμε για τα θέματα αυτά, ούτε για τα LuxLeaks προηγουμένως, ούτε για τα έγγραφα του Παναμά, ούτε για τις Μπαχάμες στην πρόσφατη αυτή δημοσίευση. Γι' αυτό σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξασφαλίστε ότι υπάρχει πραγματική και αποτελεσματική προστασία των whistleblowers, των καταγγελόντων στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλερίξ. Το τελευταίο σημείο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η προστασία αυτών που καταγγέλουν τα κακοσκήμενα, των whistleblower. Ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό στόχος. Πρέπει να βελτιωθούν η προστασία, να βελτιωθούν οι δυνατότητες προστασία των whistleblower. Αν δεν έχουν ε, προστασία τα άτομα αυτά, τα στοιχεία αυτά δεν θα γίνονταν γνωστά και δεν θα επιτύχουμε πρόοδο για πιο δίκαιη φορολόγηση. Επόμενος είναι ο Όλιβερ Τσίλμαν από την εφημερίδα Le Matin Dimanche που είναι εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορεί την Κυριακή. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Θέλω να αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν θα σας ε, δώσω περισσότερα στατιστικά στοιχεία. Ε, κάτι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Αφορά την Κύπρο και την Ελβετία. Η Κύπρος είναι δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει να είναι αντικείμενο εποπτείας από τα όργανα της Ένωσης και στα έγγραφα του Παναμά είδαμε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στα πλαίσια του κλάδου offshore στην Κύπρο. Βρήκαμε διάφορα δικηγορικά γραφεία που δρούσαν ως ε, πραγματικοί δικαιούχοι, αλλά στην πραγματικότητα έκρυβαν τους ε, ε, τελικούς δικαιούχους. Και ορισμένοι ήταν απλώς πληρεξούσιοι. Και τους βοηθούσαν Ελβετοί δικηγόροι που χρησιμοποιούσαν παραθυράκια στην ρυθμιστική διαδικασία της Ελβετίας. Ποιος το κάνει αυτό? Θέλω να σας το δείξω μια περίπτωση που θα την ξέρετε. Νομίζω. Εδώ βλέπετε δεξιά σε αυτήν την εικόνα είναι ο κ. Σεργέη Ρολντούγκεν που είναι πολύ στενός φίλος του κυρίου Πούτιν για εδώ και 40 χρόνια. Εδώ το βλέπουμε να είναι νονός του πρώτου παιδιού του κυρίου Πότιν. Ο κύριο Ρολντούκιν είναι μουσικός και δεν μοιάζει να έχει πολλά περιουσιακά στοιχεία. Το άλλο τμήμα της ιστορίας είναι ο κύριος Κόβαλτσουκ που όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είναι ο προσωπικός τραπεζίτης του κυρίου Πούτιν. Από το 2014 ε, υφίσταται, είναι αντικείμενο κυρώσεων. Του έχουν επιβληθεί κυρώσει. Η τράπεζα του κυρίου Καβαλτσούκ τι κάνει, ε, δημιουργεί μια εταιρεία offshore στον Παναμά ε, για τον κύριο Ρολντούγκιν. Τώρα γιατί ένας μουσικός χρειάζεται εταιρεία offshore στον Παναμά δεν είναι σαφές, αλλά φαίνεται ότι τη χρειάζεται. Ο κύριος Καβαλτσούκ είναι ο μεγαλύτερος ε, κάτοχος μετοχών ε, της τράπεζας της ε, Ρασίγια. Και διάφορες εταιρείες με έδρα στον, στον Παναμά έχουν λογαριασμού στην Κύπρο. Άρα τα χρήματά τους ήταν στην Κύπρο. Αλλά η Μπαν Κρασίλια ήθελε να είναι ο πραγματικός διαχειριστής αυτών των πόρων. Και για να το κάνει αυτό χωρίς να φαίνεται, χρησιμοποίησαν Ελβετούς δικηγόρους από τη Ζηρίχη. Αυτοί έκαναν όλες τις πληρωμές, αυτοί διαχειρίζονταν όλες τις εταιρείες του κυρίου Ραλντούγκιν. Αν κοιτάξετε περισσότερο τι έκαναν αυτές οι εταιρείε μέσω των εγγράφων του Παναμά, εκεί βλέπουμε ότι ο κύριος Ραλντούγκιν δεν εμφανίζεται πουθενά. Είναι σαν να μην υπάρχει στα έγγραφα, αν και είναι ο ιδιοκτήτης των εταιρεών. Και η τράπεζα του Καβαλτσούκ χρησιμοποιεί πάρα πολύ τους Ελβετούς δικηγόρους. Κάνουν πολλές ε, δοσοληψίες. Λαμβάνουν τεράστια δάνεια αυτές οι εταιρείε. Άρα τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε μια ρωσική τράπεζα στην Κύπρο. Εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμυρίων δολαρίων. Τα βλέπουμε αυτά στα γράφα του Παναμά. Κατόπιν μεταφέρονται τα χρήματα αυτά σε διάφορες ύποπτες δικαιοδοσίες όπως λένε όλοι οι εμπειρογνώμονες. Για παράδειγμα, σε ένα θέρετρο, ένα ξενοδοχείο ε, που ανήκει σε κάποιον από το στενό περιβάλλον του κυρίου Πούτιν. Σε αυτό το θέρετρο έγινε και ο γάμος της κόρης του. Επίσης κάποιες εταιρείες βλέπουμε ότι αποκτούν μυστικά δικαιώματα να ε, ελέγχουν εταιρείες που παράγουν όπλα και να αγοράζουν ε, ε, αγαθά πολυτελείας. Ε, γύρω στα δύο δις περάσανε από αυτέ τι εταιρείε του κ. Ρολντούγκιν σε διάφορα μέρη. Όλα αυτά είναι ε, ιδιαίτερα περίεργα, αφορούν δισεκατομμύρια και πολλούς γνωστούς πολιτικούς. Όλα αυτά μπορεί να είναι νόμιμα, αλλά ποιο στην πραγματικότητα αποφελείται και ποιο ελέγχει. Στην Κύπρο έχουμε μία τράπεζα είναι μια θηγατρική ρωσικής εταιρείας που ανήκει στο ρωσικό κράτος. Άρα ελέγχουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες από που προέρχονται τα χρήματα. Και επίσης έχουμε και τους δικηγόρους ε, από την Ελβετία που διαχειρίζονται αυτές τις εταιρείες και ελέγχουν τα πάντα και έχουν και την εποπτεία και με βάση τον ελβετικό νόμο τη Ελβετία και οπωσδήποτε τη Ένωση, ένα Ελβετό δικηγόρο πρέπει να κάνει τη δέουσα επιμέλεια για όλα αυτά τα οποία διαχειρίζεται, τα χρήματα που μπαίνουν στην εταιρεία του, που πάνε, από πού έρχονται και ποιο είναι ο πραγματικό δικηγόρος. Αλλά οι Ελβετοί δικηγόροι χρησιμοποιούν μια δυνατότητα, μια ευκαιρία που του προσφέρει η Μοσάκ Φοντσέκα. Είναι οι λεγόμενοι δικαιούχοι διευθυντές ή ορισμένοι διευθυντές οι οποίοι στην ουσία είναι βιτρίνα, υπογράφουν τα πάντα χωρίς να διαχειρίζονται. Υπάρχει ένα παραθυράκι στο ελβετικό δίκαιο που, λένε ότι, που λέει ότι αν δεν υπογράφει εσύ για μια εταιρεία δεν χρειάζεται να κάνει τη δέωση επιμέλεια. Δηλαδή οι δικηγόροι στην Ελβετία μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν χρειάζεται να εξετάζουν τακτικά πώς λειτουργούν και τι δοσοληψίες κάνουν αυτές οι εταιρείες. Τελικά θα έπρεπε βέβαια να ελέγχουν ε, οι αρχές του Παναμά γιατί θεωρητικά είναι υπεύθυνοι. Μια που εκεί στον Παναμά είναι η αυτοί οι εικονικοί διευθυντές. Ρωτήσαμε τις αρχές του Παναμά. Εξετάσατε αυτά τα άτομα. Είναι άτομο του στενού περιβάλλοντος του κ. Πούτιν, ο κ. Ροντούκιν. Και η γραπτή τους απάντηση είναι ότι έχουμε μια πολύ γνωστή και έγκυρη ε, εταιρεία δικηγόρων στο, στην Ελβετία η οποία θα πρέπει να ελέγχει. λέει τι μας λένε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα εμείς. Οι Ελβετοί πρέπει να τα κοιτάξουν. Διότι οι Ελβετοί έχουν τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες τις οποίες δεν ασκούσαν. Άρα κανείς δεν έλεγχε. Στην ουσία είναι μια δομή η οποία αξιοποιεί τα παραθυράκια. Εδώ πρέπει να εξετάσουμε γιατί με αυτή τη δομή ήταν δυνατόν άτομα του στενού περιβάλλοντος του κυρίου Πούτιν να περάσει εκατοντάδες εκατομμυρίων δάνεια χωρίς έλεγχο μέσω δικαιοδοσιών της Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρόνο σας. Τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία ε, Στάιν και τον κύριο Στρότσι. Παρακαλώ, πέραστε. Εδώ στο, στην έδρα. Καλώ äh, Καλώς ε, ήρθατε κυρία Στάιν και στο κύριο Στρότζεκ τον ε, καλωσορίζω από, την, από το ραδιόφωνο της Βόρειας Γερμανίας στο Αμβούργο στην Γερμανία. Έχετε το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση και την ευκαιρία να μπορέσω να λάβω το λόγο ενώπιον της Επιτροπής σας σαν Επιτροπή Ερεύνης, εσείς προφανώς ερευνάτε παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου, Δικαίου και παραλήψη της Κομισιόν, αλλά βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολο, ακόμα και σε όταν, όταν πρόκειται για τόσο μεγάλες διαρροές εγγράφων, να κατανοήσει κανείς και να αποδείξει ότι υπήρξαν παραβιάσεις του δικαίου. Συνήθω έχουμε έλλειψη των αποφασιστικών στοιχείων πληροφορία που καταδεικνύει ότι υπήρξε μια παραβίαση του φορολογικού δικαίου και βοηθούν τι φορολογικέ και διοκτικέ αρχέ. Το να, το να μπορέσουμε όμω να αποδείξουμε ότι υπήρξαν κάποιε παραβιάσεις το καταφέραμε με τα Panama Papers. Παραδείγματο χάρη υπήρξε μια παραβίαση από την πλευρά τη εταιρεία Mossack Fonseca όταν ο Ράμι Μαχλούφ, ο οποίο ήταν ο ξάδερφος του Μπασάρα Λασάντ, ε, είχε, είχε φανεί ότι ήταν πελάτη. Ενώ αυτό έρχεται σε σύγκρουση με τι συγκρούσει. Υπάρχουν λοιπόν και άλλοι εγκληματίες που φαίνονται στα Panama Papers, οι οποίοι λειτουργούν ως πελάτες για να κρύψουν την περιουσία τους και αυτό είναι πάλι σαφής παραβίαση του δικαίου. Το να εξασφαλίσουμε βέβαια ότι κάποιος τους έχει αρρωγήσει σε αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. <clears throat> Πέραν αυτών των συγκεκριμένων παραβιάσεων που ανέφερα προηγουμένω, εμένα με ενοχλεί περισσότερο το ότι υπάρχει μια συστηματική λειτουργία πίσω από αυτά. Γιατί υπάρχει η νομική δυνατότητα και είναι νόμιμο να έχει κανείς μια εταιρεία ε, γραμματοκιβατίου. Και αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα αφ' αυτού. Μπορεί κανείς να έχει και μια τέτοια εταιρεία την οποία την πωλεί σε κάποιον άλλον. Είναι επίσης ε, νόμιμο να ζητά κανείς να δώσει σε κάποιον τη δυνατότητα να είναι ο δικαιούχος ε, μιας εταιρείας η οποία όμως τον, του επιτρέπει να παραμείνει ανώνυμος. Με τον τρόπο αυτό δεν μπορεί κανείς ποτέ να ελέξει τι είναι νόμιμο και τι δεν είναι νόμιμο γιατί υπάρχει αυτή η απόλυτη αδιαφάνεια πολλοί είναι αυτοί σε στο, στο παγκόσμιο στερέμα που θέλουν να έχουν τέτοιε εταιρείε γραμματοκιβωτίου. Είναι η κορφή του παγόβουνου, η μύτη του παγόβουνου μονάχα η Μοσάκ Φονσέκα και ο Παναμά είναι μονάχα μία από διάφορε φορολογικέ οάσει στον κόσμο. Και πολλές τράπεζες έχουν ε, γραφεία και θηγατικές που εξυπηρετούν αυτή τη διαδικασία. Αν δείτε λοιπόν στο ίντερνετ πώς μπορείτε να φτιάξετε μια απο διάφορε φορολογικέ οάσει θα δείτε πολλέ τράπεζε εχουν μεγάλο κατάλογο ε, ευκαιριών που εξυπηρετουν αυτη τη διαδικασια αν δειτε λοιπον στο ιντερνετ πώ μπορειτε να φτιαξετε μια εταιρεια γραμματοκιβωτιου θα δειτε ενα πολυ μεγαλο καταλογο ευκαιριων που δινει που παρουσιάζονται στο διαδίκτυο. Και αναρωτιέται κανείς ε, ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση για αυτές τις εταιρείε. Λένε όλες αυτές στο διαδίκτυο ότι θα σας δώσουν απόλυτη εμπιστευτικότητα. Υπάρχει υψηλό επίπεδο ανωνυμίας και προστασίας της προσωπικής σας ζωής. Αυτό σας υπόσχονται. Και λένε επίσης και παραθέτω ότι δεν θα πληρώσετε κανένα φόρο οποιοδήποτε είδους. Αλλά πιο γνωστό από όλα είναι το γεγονός ότι ο Παναμάς είναι μια χώρα που έχει μια πολύ καλή ε, φήμη μέχρι βέβαια την ε, ανακάλυψη των Panama Papers. Όλες αυτές λοιπόν οι επιχειρήσεις ουσιαστικά έχουν ένα σκοπό να βοηθήσουν άλλους να φτιάξουν εταιρείε γραμματοκιβωτίου. Απλώς αρκεί να έχει κανείς μια ε, διεύθυνση email και ένα διαβατήριο και με, με λίγα κλικ μπορεί κανείς να εξασφαλίσει ότι θα γίνει ο ιδιοκτήτης μιας ε, εταιρεία, είτε οι δουλειές του είναι νόμιμες είτε είναι παράνομες, δεν πρόκειται να κινδυνεύει να τον ελέγξει κανείς. Η τεκμηρίωσή μας για την ε, ταινία που παρουσιάσαμε και το ντοκιμαντέρ που παρουσιάσαμε στην NDR-RD είχαμε αναφερθεί σε μία σειρά από εταιρείες οι οποίες ε, έχουν έδρα στο Παναμά. Ο εισηγητής μας, ο Κρίστοφ Λίτκερτ, έχει παρουσιάσει τώρα ένα βίντεο το οποίο ελπίζω θα μπορέσετε να δείτε και θα σας δείξει τι καταφέραμε να πετύχουμε να βρούμε μέσω των εγγράφων του Παναμά. Gut, solange es nicht funktioniert, kann ich versuchen es. Επειδή δεν λειτουργεί, να σας ε, περιγράψω κάπως την κατάσταση. Ε, μου είχατε πει ότι έχετε ίντερνετ. Ε. Φαίνεται πως δεν έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίντερνετ. Προσπαθήσαμε να παρακολουθήσουμε την, να βρούμε ποια ήταν η διεύθυνση. Πήγαμε λοιπόν στη διεύθυνση αυτή. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα κτίριο. Δεν ήταν εύκολο να μπούμε να δούμε τα γραφεία. Πήγαμε στο 19ο όροφο. Γιατί στο 19ο όροφο όμως, όταν φτάσαμε, είδαμε ότι ήταν για πει το κτίριο. Στο ίντερνετ διαπιστώσαμε ότι στην ίδια διεύθυνση έχουν έδρα 6.000 εταιρείε. 6.000 εταιρείε έχουν έδρα ένα για γιαπί. Όταν το είδαμε καταλάβαμε πόσο παράλογο είναι ε, το όλο σύστημα. Ε, με λίγα κλικ, χωρίς να μιλήσεις με κανένα, στην ανωνυμία του ίντερνετ, ε, ξαφνικά γίνεσαι ιδιοκτήτης εταιρεία. Πώς είναι δυνατόν να είναι νόμο κάτι τέτοιο. Πώς είναι δυνατόν να διαφημίζουν στο ίντερνετ εταιρείε ε, των οποίων ο ιδιοκτήτη θα είναι απόλυτα ανώνυμο. Πώ δυνατόν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Ακόμη και αν υπάρχει ένα μητρό όπου αναφέρονται οι εξοδοτημένοι, πάρα πολλά ξεφεύγουν. Πότε θα έχουμε παγκόσμιε προδιαγραφέ για το τι πρέπει να δηλώνεται, πότε θα είναι συνδεδεμένα όλα αυτά. Χρειαζόμαστε να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο επιγόντω. Εάν ε, πιέσει περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κερδίσουμε πολλά. Αυτή τη στιγμή αρχές όλο τον κόσμο προσπαθούν να διαλευκάνουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις και στη Γερμανία. Οι αρχές ε, της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας προσπαθούν να αποκτήσουν την πληροφόρηση για όλα αυτά τα στοιχεία και έχουμε ήδη ε, έρευνες για 400 τέτοιες εταιρείες. Υπάρχουν επίσης έρευνες σε διάφορα άλλα ομόσμοδα κράτη. Και επίσης οι γερμανικές τράπεζες όλο και περισσότερο είναι στο στόχαστρο. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ε, το φιλμ ακόμη δεν μπορούμε να το δείξουμε. Εν πάση περιπτώσει μπορείτε να το δείτε στο ίντερνετ και μπορείτε να δείτε ότι πρόκειται για γιαπή πραγματικά. Ο κύριος Στρότσικ. Ευχαριστώ Γιούλια. Κυρίες και κύριοι. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να συνεχίσω με αυτά που είπε η Γιούλια τι ρόλο δηλαδή παίζουν οι ενδιάμεσοι και τι μπορεί να επιτύχει κανείς μέσω της ε, Μοσάκ Φονσέκα. Γιατί λοιπόν πρέπει να ασχολούμεθα εμείς με μια δικηγορική εταιρεία στον, στο Παναμά. Αυτό το κάνουμε εμείς ως δημοσιογράφοι, διότι Ορισμένες από τις παρανομίες γίνονται εδώ στην Ευρώπη. Πρέπει να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Η Μοσάκ Φονσέκα, όπως ε, πολλοί άλλοι οι οποίοι προσφέρουν offshore εταιρείε δεν έρχονται σε επαφή απευθείας με τον τελικό πελάτη. Υπάρχουν διάφοροι ενδιάμεσοι, intermediaries. όπως λέει και το όνομά τους, ε, είναι ανάμεσα στην Μοσάκ Φονσέκα και τον τελικό πελάτη. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί η Μοσάκ ε, Φονσέκα είναι σαφές και συχνά μας το ανέφεραν, για να μπορούν να μας πούνε εμείς δεν έχουμε καμία επαφή με αυτόν τον πελάτη. Πάντα μπορούν να μας ε, πούν κάτι τέτοιο, να κάνουν αυτόν τον ισχυρισμό. Now Καλώς συνεχίζει ο κύριος Στρότσεκ μετά από τη διακοπή είναι και μια μορφή ε, ε, από, ε, μεταφορά σε άλλον της ευθύνης. Στην ουσία αυτό λέγεται μεταφορά της ευθύνης για την δέουσα επιμέλεια σε κάποιον άλλον. Δηλαδή στην ουσία κάποιοι ενδιάμεση λένε ότι τα πράγματα είναι καλά και η Μωσά Φωνσέκα λέει εντάξει το πιστεύω. Είναι μεταφορά λοιπόν ευθύνη. Στην ουσία δηλαδή ε, δεν είναι σαφές και ποια ε, ρυθμιστική αρχή έχει την ευθύνη. Και αυτό είναι το μοντέλο. Μοσάκ Φονσέκα ως δικηγορικό γραφείο στον Παναμά ποτέ δεν θα έχει δυνατότητα να εξυπηρετήσει τόσους πελάτες. Οι πλούσιοι πελάτες των εταιριών στην ουσία προσανατολίζονται από τις τράπεζες προς τέτοιες εταιρείες ούτως ώστε να υπάρχουν λιγότερες ε, λιγότερα ίχνη για το τι γίνεται. Εγώ πηγαίνω στην τράπεζα, συζητώ με τον σύμβουλό μου, με τον οποίο εργάζομαι πολλά χρόνια και τον ε, ε, εμπιστεύομαι και κατόπιν ε, συμφωνούμε πού θα ιδρυθεί αυτή η εταιρεία γραμματοκιβώτιο ούτω ώστε να μπορεί αυτό το άτομο να πει μετά, εάν ρωτηθεί, ότι η εταιρεία αυτή δεν είναι δική του. Όλα αυτά τα είδαμε στα έγγραφα, όλα αυτά γίνονται με πολύ επαγγελματικό τρόπο. Υπάρχουν ε, ήδη έγγραφα τα οποία έχουν συμπληρωθεί χωρίς να έχουν υπογραφεί και υπάρχει και ανταλλαγή υπαλλήλων, δηλαδή αποσπώνται από τη Μοσάκ Φονσέκα σε τράπεζες και αντίστροφα. Δηλαδή πα σε κάποιον και σου παρέχει ό,τι υπηρεσίες θέλεις. Είχαμε ε, βρει και άλλα έγγραφα πριν από τις διαρροές του Παναμά και εκεί είχαμε διαπιστώσει ότι ισχύει το ίδιο μοντέλο. Από τις 7 μεγαλύτερες γερμανικές τράπεζες, οι 6, όπως είδαμε από τα έγγραφα του Παναμά, είχαν οργανώσει ή διαχειρίζονταν εταιρείε για τους ε, πελάτες τους με μεγάλο ε, όγκο περιουσιακών στοιχείων. Και αν εξετάσουμε και τα προηγούμενα στοιχεία που είχαμε, διαπιστώνουμε ότι από τις 20 μεγαλύτερες θράπεζες του κόσμου, οι 13 ε, εμφανίζονται μέσω όλων αυτών των διαρροών να έχουν τέτοιες εταιρείες. Δεν είναι όμως μόνο ότι απλώς προσφέρουν τέτοιες εταιρείες γραμματοκιβωτίων, στους πελάτες τους για να τους εξυπηρετήσουν βγάζουν χρήματα από αυτές τις επιχειρήσεις και σε άλλες χώρες όπως το Λουξεμβούργο και η Ελβετία όπως υπόθηκε ορισμένες ε, τράπεζες που έχουν εμπλακεί στην Γερμανία είναι τράπεζες όπου συμμετέχει το κράτος ως ε, ε, μέτοχος ή που έχουν διασωθεί μέσω κρατικών πόρων. Υπάρχουν ε, και άλλοι που συμμετέχουν, είναι πάρα πολλοί δικηγόροι, διάφοροι που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία. Είναι μια αγορά που δεν υπόκειται σε πολλές ρυθμίσεις. Διάφοροι ιδιωτικά αυτοαπασχολούμενοι με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, πολλοί που είναι γνωστοί των ανθρώπων με μεγάλη περιουσία. Δεν θα τα αναφέρω όλα αυτά γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει νομίζω να εστιάσουμε περισσότερο στις τράπεζες γιατί οι τράπεζες είναι πολύ πιο συστημικό στοιχείο όλη αυτή τη ε, διαδικασία. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι αναλαμβάνουν όλες υπηρεσίε υπηρεσίες, ε, one-stop shop, οι οποίοι εργάζονται με πολύ τελειοποιημένο τρόπο. Και επίσης συμμετέχουν βέβαια και οι μεγάλοι τέσσερις σύμβουλοι, οι τέσσερις μεγάλες εταιρείες ε, λογιστικού ελέγχου και παροχής συμβουλών. Προσπαθούμε να βρούμε κάποια στοιχεία. Στα έγγραφα του Παναμά αναφέρονται πάνω από 500 τράπεζες. 30 έχουν σχέση με τη Γερμανία. Είναι είτε γερμανικές τράπεζες που έχουν έδρα στη Γερμανία, που έχουν και δραστηριότητα στο εξωτερικό ή τράπεζες που έχουν έδρα στο εξωτερικό αλλά που έχουν δραστηριότητα και στη Γερμανία. Από τις πιο σημαντικές 10 τράπεζες που παίζουν ρόλο ενδιάμεσου τέσσερις από το Λουξεμβούργο, τρεις από ε, νησιά της Καραϊβικής, δύο από το Λουξεμβούργο και μία από την Ελβετία. Άρα είναι τράπεζες που σε όλες μπορεί να πας ε, γρήγορα, με κάποιες ώρες της. Ένας ε, συνεργάτης της Μοσάκ Φονσέκα στο Λουξεμβούργο μας είπε ότι δεν θα έπρεπε να σας εκπλήσει το ότι οι δουλειές μας πάνε θαυμάσια. Σε μία ε, συγκεκριμένη εβδομάδα μας είπε ότι είχε δημιουργήσει και πωλήσει 115 εταιρείε γραμματοκιβώτιο. Ένα μόνο γραφείο στο Λουξεμβούργο, όχι στον Παναμά, όχι στις Μπαχάμες, όχι μακριά. Αυτές οι συναλλαγές γίνονται εδώ, ανάμεσά μας. Είναι σημαντικό στοιχείο. Οι συνάδελφοι αυτού του μου δημοσιογράφων έχουν κάνει μια πολύ ωραία παρουσίαση όπου συνοψίζουν ποιοι είναι οι ενδιάμεσοι που βλέπουμε που διαπιστώσαμε μέσω των διαρροών του, των Μπαχαμών και του Παναμά είναι 24.000 και παραπάνω. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση όταν μας ρωτάτε με ποιους, σε ποιους μπορούμε να απευθυνθούμε. Έχετε αυτό το κατάλογο, μπορείτε να διαβάσετε αυτό το κατάλογο για να δείτε ποιους μπορείτε να προσκαλέσετε από όλους αυτούς τους ενδιάμεσους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στρότσερ και κυρία Στάν και θα δώσω το λόγο στην κυρία Κνούτ. Κνούτ, συγγνώμη. Καλώ ήρθατε κυρία Μίνα Κνού, από την ε, Φιλανδική Ραδιοτηλεόραση. Στα έγγραφα ε, που σας έχουν διανυμηθεί βλέπετε και τα βιογραφικά όλων των δημοσιογράφων, άρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερη παρουσίαση. Κυρία Κνούς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Είναι τιμή μου. Έχω ένα λεπτομερέστατο έγγραφο, αλλά θα προσπαθήσω να συνοψίσω τις βασικές ιδέες αυτή τη σύντομη παρουσίαση. Έχω χωρίς, ελπίζω να δουλεύει αυτό. Πού πατάω, πού δείχνω. Α, εκεί, ωραία. Έχω χωρίσει τα ευρήματά μας από τη Φινλανδία σε τέσσερις ομάδες. Νομίζω οι σημαντικότερε ομάδε που θα, θα πρέπει να σα αποσχολήσουν, όπω είπαν και κάποιοι από του συναδέλφου μου, είναι οι μεσάζοντε, οι δύο τράπεζε. Διότι εκεί ήταν ο καλά οργανωμένο σε επίπεδο κλαδικό τρόπο για να δημιουργούνται εταιρείε offshore, εταιρείε φαντάσματα. Οι βασικέ υποθέσει στην Φιλανδία ήταν η Νορντέα και Μέτσο στις οποίες εν μέρει η ιδιοκτήτης είναι το κράτος το ίδιο της Φιλανδίας. τα ευρήματα από την Ορντέα. 400 εταιρείε offshore, μόνο και μόνο από το αποκατάστημα Ορντέα του Λουξεμβούργου. Υπήρχαν και offshore εταιρείε από την Ελβετία, αλλά εντοπίστηκαν κυρίω από το Λουξεμβούργο στον Παναμά και μερικέ στι νήσου τη Παρθένου. Ξέρετε βεβαίω για τη Μοσάδο Φονσέκα και Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η ανάμειξή του, Ο πελάτης είναι μεσάζων στον κόσμο, στο σύμπαν αυτό της ε, Μοσάκ Φονσέκα. Με πολλές τρώσει μυστικότητα, όπως ε, ανώνυμους μετόχους, ε, με αναπληρωτέ διευθυντέ, με ιδρύματα. Βρήκαμε Και αυτό είναι μέρο ενό email από το υποκατάστημα τη Νορδέας στο Λουξεμβούργο προ τη Μουσάκη Φωνσέκα που λέει διαγράψτε το όνομα αυτού του αναπληρωτή διευθυντή, μάλλον αυτή τη αναπληρωτή διευθυντή, γιατί έχει πεθάρει εδώ και 8 χρόνια. Διαγράψτε το από όλα τα έγγραφα ή τέλο πάντων αλλάξτε το όνομα. Αυτό το έγγραφο είναι το 2008 και η αναπληρώτρια διευθύντρια πέθανε το 2005. Το έγγραφο δεν έχει καμία σχέση με την Ορντέα. Είναι όμως, είναι, δείχνει πόσο παράλογο είναι το σύστημα αυτών των αναπληρωτών διευθυντών. των πληρεξούσεων μάλλον διευθυντών. Βρήκαμε πολλά έγγραφα ετεροχρονισμένα. Η Νορντέα ε, ζήτησε να πάει ένα έγγραφο μία διετία πίσω για έναν ε, εταιρικό δικηγόρο και βεβαίω ο Ζακ Φονσέκα είπε κανένα πρόβλημα αρκεί να πληρώσετε. Για ένα χρόνο ετεροχρονισμένο εγγράφο 200 δολάρια, για δύο χρόνια 350. Αυτέ ήταν οι αμοιβέ τους. Η περίπτωση τη Νορντέα ήταν αποτέλεσμα ε, δημοσιογραφικής συνεργασίας με σκανδιναβούς συναδέλφους οι οποίοι ε, βρήκαν πολλά σκιαδάνια και υπήρξαν πολλές ενδιαφέρουσες συναντήσεις με λεπτομερή σχόλια από τις συζητήσει μας με τους υπευθύνους της Μοζακονσέκα και της Νορντέα. Αν δείτε ότι πραγματικά είναι ένα παιχνίδι της ε, ποντικοπαγίδας εδώ. Ε, όταν έρχεται κάποιος καινούριο πελάτης, ψάχνουν καινούριε λύσεις, ψάχνουν ε, και αγρεύουν νέα δικαιοδοσία. Βλέπουμε εδώ ότι η υπόθεση Panama Papers αποδεικνύει ότι όσα συνέβησαν στο Λουξεμβούργο συνεχίστηκαν παρά τις προειδοποίησεις. Η Νορντέα είχε λάβει προειδοποίησεις επανειλημμένως από τις σουηδικές ε, ε, φορολογικές αρχές λόγω της περίπτωσης του Λουξεμβούργου και της πολύ κακής αντιμετώπισης του θέματος ε, ξεπλήματος βρωμικού χρήματος και τελικά δεν το έλαβαν επαρκώς υπόψη τους. Η άλλη περίπτωση είναι η Μέτσο, μια μεγάλη εταιρεία της Φινλανδίας, στην οποία έχει μεγάλη συμμετοχή και το Φινλανδικό κράτος. Ήταν μια περίπτωση ξεκάθαρη ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, και ε, ο διευθυντής της Μέτσο από τη Ρωσία μπορούσε να προωθεί το χρήμα από τη δική του ε, ιονή εταιρεία στον Παναμά μέσω της Μέτσο. Δηλαδή πλήρωνε από τη δική του εταιρεία φάντασμα του Παναμά με τον ελβετικό του λογαριασμό στην Ορντέα στο Ελσίνκι και τα ίδια προϊόντα πολλούνταν σε σουηδική εταιρεία, αλλά έξι φορέ ε, πάνω από την τιμή του. Αυτό το παραπάνω χρήμα πήγαινε σε μια βρετανική εταιρεία και πίσω στι τσέπε του διευθυντή αυτού στην εταιρεία Φάντασμα στον Παναμά. Αυτό κατέστη εφικτό χάρη σε αυτές τις ανώνυμες εταιρείες, τις κενές ε, κατά τα άλλα εταιρείες, με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, χρυσό, πολύτιμα ε, μέταλλα, με την εταιρεία που ε, έχει δημιουργήσει Mossack Fonseca για να χειρίζεται τέτοια ποσά και περιουσιακά στοιχεία. Κι άλλη στρώση μυστικότητα αυτή, γιατί κανεί δεν μπορεί να δει ποιο χειριστατέ χρηματοοικονομικέ συναλλαγέ. Η φιλανδική αστυνομία δεν μπορεί ακόμη να κάνει έρευνα για, την, ε, για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο από τη Μόσα Φονσέκα, ε, γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι υπεύθυνο, παρόλο που τόσε ευρωπαϊκέ χώρε είναι μπλεγμένε στην υπόθεση. Μπορεί να συνεχίσει λοιπόν ανενόχλητο και να συνεχίσει με τι σουηδικέ του και ελβετικέ του εταιρείε ο άνθρωπο αυτό. Ε, και εδώ. Και ήθελα να σα το πω αυτό γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Έχουμε μια δικαστική υπόθεση στη Φιλανδία. Οι φιλανδικέ ε, φορολογικέ αρχέ θέλουν τα στοιχεία από τη δική μας συντακτική έρευνα, τη δημοσιογραφική έρευνα και τα πορίσματά μας. Είναι πολύ επιθετικές φορολογικές αρχές. Δεν ξέρω καμία άλλη χώρα όπου οι δημοσιογράφοι που ασχολήθηκαν με το όλη προσπάθεια Panama Papers να βρέθηκαν σε αυτή τη θέση. Είπαμε βεβαίω όχι, δεν μπορούμε να σας δώσουμε ούτε την ερευνά μας, ούτε τα πορίσματα υπόθεση ακόμα εκδικάζεται σε διοικητικό δικαστήριο του Ελσίνκη και θα τραβήξει η βαλίτσα. Οι δικηγόροι λένε ότι η πρώτη απόφαση μπορεί να βγει το επόμενο καλοκαίρι. Α, θα σκίσουμε έφεση, θα κρατήσει κι άλλο. Είναι πολύ ενδιαφέρον διότι η Φινλανδία είναι πρώτη στην ελευθερία του τύπου παγκοσμίω και έχουμε πολύ καλή προστασία των πηγών μας ως τώρα. Αυτό λοιπόν πρέπει να παρακολουθηθεί. Η ερευνητική δημοσιογραφία, ο τρόπος που χρησιμοποιούμε του πληροφοριοδότες, τις διαρροές και τις πηγές μας είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πολύ πολύ σοβαρά. Αυτά και για να ολοκληρώσω κάποια διδάγματα ίσως από αυτή την υπόθεση. Πρέπει κανείς να ψάξει το θέμα των πελατών, των μεσαζόντων, της διαφάνειας ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Είναι τόσε πολλέ οι στρώσει μυστικότητα εδώ σε αυτόν τον κόσμο των επιχειρήσεων και όλα τα μητρώα επιχειρήσεων θα έπρεπε να είναι διαφανή σε όλο τον κόσμο. Επίση, η δικαστική υπόθεση κατά των απλευροειδετών του LuxLeaks και ε, δημοσιογράφων είναι πραγματικά όνειρο αυτό για την Ευρώπη. Πρέπει να υπάρξει μεγάλη συνεργασία μεταξύ όλων στην Ευρώπη για να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδου υποθέσει που μα ντροπιάζουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κνούς. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ε, παρουσιάσεις και τις προτάσεις που μας δώσατε. Έχουμε καθυστερήσει και στο πρόγραμμά μας. Ξεκινήσαμε η αλήθεια είναι λίγο αργότερα. Ελπίζω παρόλα αυτά ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε πλήρως τον γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. Έχουμε δύο συνεισηγητές στο Ευρωκοινοβούλιο ο κύριος Γιάπο Κόφουτ από τους σοσιαλδημοκρατές της Δανία και ο Πέτερ Γέτσεκ από την Άλντε στην Τσεχία, φιλελεύθερη. Και οι δύο εισηγητές τώρα θα λάβουν το λόγο για πέντε λεπτά το πολύ. Παρακαλώ κύριε Κόφουτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους καλεσμένους μας σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεδρίαση για την Επιτροπή μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημοσιογράφους και βέβαια όλους τους whistleblowers, τους καταγγέλλοντες για την <clears throat> εργασία τους στα πλαίσια των Panama Papers. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σκοτεινός κόσμος όπου γίνονται ε, δοσοληψίες οι οποίες είναι εξοργιστικού χαρακτήρα τα χρήματα των πλουσίων χρησιμοποιούνται για να παρακάμψουν τις φορολογικές αρχές, για να, για να βοηθήσουν την τρομοκρατία, για να υποστηρίξουν ε, αυτοκρατικούς ηγέτες όπως είναι ο Ασάντ ή ο Πούτιν. Επομένως το πραγματικό ερώτημα το οποίο θέλουμε να θέσουμε όλοι γιατί πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα και να ξεπεράσουμε αυτό το επίπεδο αδιαφάνειας <clears throat> το ερώτημα προς εσάς που θέλω να θέσω είναι το εξή. Βλέπετε κάποιο νομικό εμπόδιο ή βρήκατε νομικά εμπόδια ή πολιτικά, πολιτικές πιέσεις που εμπόδισαν το έργο σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδαμε την περίπτωση αυτή του, της δικαστικής δίωξης των καταγγελόντων στο Λουξεμβούργο. Ποιε νομοθετικές πρόνοιες θέλετε να αλλάξουν στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και του ξεπλήματος χρηματών. Θα ήθελα να μπορέσετε εσείς ως δημοσιογράφοι να μας πείτε για κάτι παραπάνω για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ποιο θα ήθελε να δώσει απαντήσεις από τους δημοσιογράφους, λέει ο πρόεδρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για τα νομικά εμπόδια και την πίεση νομική. Για το Βέλγιο μόνο μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω εξ όλων των συναδέλφων από τον κόσμο. Θα γνωρίζετε ότι η ελευθερία των μέσων είναι κάτι το πολύτιμο Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα καλή προστασίας των πηγών και της ε, ελευθερία έκφρασης. Δεν έχουμε πραγματικά εμπόδια, ούτε δεχόμαστε πολιτικές πιέσεις. Ωστόσο, δικηγόροι προσπάθησαν να μας πείσουν να μην δημοσιεύσουν άρθρα για συγκεκριμένου λόγους, αλλά όπως είπαν συνάδελφοι και από άλλα μέρη του κόσμου και από άλλε χώρε με λιγότερο α πούμε δημοκρατική παράδοση, Καμιά φορά η δουλειά μας είναι δύσκολη. Ευχαριστούμε κύριε Κόφοντ. Και εσείς μπορείτε να προσθέσετε ερώτηση. Ναι, θα ήθελα να μου πει κάποιος δοσμογράφος ε, ποια είναι η νομοθεσία που θα θέλατε να αλλάξει για την ε, προστασία των μέσων. Είναι σημαντικό για μας αυτό. Είδαμε την υπόθεση των μεσαζόντων, των ε, ενδιάμεσων. Πώ θα έπρεπε να το προσεγγίσουμε εμεί αυτό κατά την άποψή σα, Τι ε, έχετε βρει στα πορίσματά σα που θα μπορούσε να μα βοηθήσει να προχωρήσουμε στη δουλειά μα στο Panama Papers. Ε, γι' αυτό είχε μιλήσει η κυρία Στάιν. Πώ θέλει να απαντήσει από αυτού. Ναι, κοιτάξτε, ο διάβολο είναι πάντα στι λεπτομέρειε και το να είναι κανεί πολύ συγκεκριμένο είναι δύσκολο. Αλλά το βασικό είναι ο τρόπο λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων. Ο τρόπο λειτουργία επιτρέπει να παραμένει ανώνυμος ο τελικός δικαιούχος. Και αυτό είναι νόμιμο. Πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει παράνομο για να μπορούμε να αποδείξουμε ότι κάνει κάτι παράνομο. Και ακριβώς, εάν δεν μπορούμε να δούμε συνολικά την αλυσίδα ε, ιδιοκτησίας και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων δεν μπορεί να ελέγξει. Και γι' αυτό τελικά χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία των γραμματοκιβωτίων για παράνομες δραστηριότητες. Και άλλε μπορεί να είναι παράνομε, άλλε να είναι εντελώ ε, νόμιμε. Χωρί μικρόφωνο μιλάει κάποιο. Παρακαλώ. Πολύ σύντομο, τελευταία ερώτηση. Καλώ αναφέρατε περισσότεροι από εσά τι τράπεζε στην Ευρώπη, όλο ιδιαίτερο. Θα ήθελα, εάν μπορείτε, να μα εξηγήσετε πόσο συνεργάζονται οι τράπεζε και οι υπευθυνοί του στην Ευρώπη για τα πορέσματά σα και στη δουλειά σα ω δημοσιογράφων. Ω μεσάζοντε, οι τράπεζε έχουν και αυτέ ευθύνε, προφανώ. Τι εμπόδια έχετε εντοπίσει, Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να αναγκαστούν να συνεργάζονται καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ποιο θέλει να απαντήσει, Η κυρία Κλού. Α, όχι. Στην ε, περίπτωση της Νορντέα, ο αντίκτυπος της σκανδιναβικής χώρας ήταν τεράστιος με την Νορντέα. Στη Φιλανδία είναι μπλεγμένα πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ιδιώτες, φύγαν. Κλείσαν τους λογαριασμούς τους από την Νορντέα, κανονικά. Η Νορντέα λοιπόν χρειάστηκε να το πάρει πολύ σοβαρά υπόψη αυτό που γινόταν. Έγινε ολόκληρη έρευνα μετά στο Λουξεμβούργο. Νομίζω ότι η δημοσιότητα πραγματικά έκανε μεγάλη διαφορά. Τους ανάγκασαν να το δουν πολύ σοβαρά. Προηγουμένως η συνεργασία μας, σε συνεντεύξεις που είχαμε μαζί του και συνομιλίε ήταν κάπως δύσκολες. Όταν ήταν, είδαν πόσο πολύ επηρέασε το κοινό, πόσο θύμωσε ο κόσμος, τότε κατάλαβαν ότι πρέπει να το πάρουν σοβαρά. Το παίρνουν πολύ σοβαρά πλέον στη Φιλανδία. εκτός μικροφώνου. Απλώς να προσθέσω από την προοπτική της Ελβετίας που έχει και τα πάει καλά με τράπεζες. Εμείς μετατοπιστήκαμε λίγο στη χώρα μας, αν το δείτε από την άποψη των τραπεζών. Δηλαδή, ενώ προηγουμένως περισσότερες εταιρείες offshore το 2005 ως ήταν ένα μέσο για να κατευθύνει κανείς τις οικονομίες του, τις εξοικονομήσεις του, τις κατεύθυνε από την Ελβετία προς το εξωτερικό και εκεί αναλάμβαναν δικηγόροι. Βλέπουμε ότι η τάση ήταν να αναλάβουν καθαρά, σκέτο, ε, καθαρά τα δικηγορικά γραφεία που έχουν λιγότερη εμπειρία από τις τράπεζες. Τους δικηγόρους σας μεσάρτες πρέπει να δείτε λοιπόν. Ευχαριστώ. Ο Πέτερ Γέτσεκ, ο άλλος συνεισηγητής, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ όλους τους δημοσιογράφους που πήραν το λόγο και να τους συγχαρώ επίσης για το ότι τήρησαν το χρόνο και έδειξαν ε, ότι είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμοι. Θαυμάσια ομαδική εργασία. Θα ήθελα τη γνώμη σας για τα εξή θέματα. Πρώτα απ' όλα, ποιες είναι οι διαστάσεις του προβλήματος, τα έγγραφα του Παναμά και οι άλλε αποκαλύψει Είπατε ότι είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ποια είναι η διάσταση, η πραγματική του προβλήματος. Δεν θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε και άλλες διαρροές επί των οποίων εργάζεστε, αλλά τι άλλο μπορείτε να μας πείτε. Και όλα αυτά τα μοντέλα φοροδιαφυγής. Από ό,τι κατάλαβα, ανεξάρτητα από το σε ποια χώρα είναι, είναι περίπου τέτοια τα σχήματα με ενδιάμεσου, με εταιρείε προπετάσματα κτλ. Κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό είναι γιατί προκύπτουν αυτά τα θέματα. Ποια είναι τα κύρια εμπόδια για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Γιατί παγκόσμια δεν έχει υπάρξει πολύ περισσότερη πρόοδος, πολύ πιο ουσιώδης πρόοδος. Γιατί οι κυβερνήσεις της Ευρώπης δεν το θεωρούν προτεραιότητα. Γιατί γιατί είναι ανίκανες να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το θέμα των φορολογικών ε, παραδείσων ή η νομοθεσία δεν επαρκεί. Η κυρία Στάιν τόνισε ήδη ότι η ουσία του προβλήματος είναι αυτές οι εταιρείε προπέτασμα, η ανωνυμία τους και το γεγονός ότι είναι νόμιμες παρόλα αυτά ότι θα έπρεπε λοιπόν, είπε, ε, κατά πάσα πιθανότητα να βελτιώσουμε την νομοθεσία. Και για το μέλλον, πώς θα διασφαλίσουμε την εφαρμογή των συστάσεών μας. Θα συνεχιστεί η πίεση των μέσων επί των κυβερνήσεων και σε εμά και εφημών. Διότι υπάρχουν και διάφορες κυβερνήσεις οι οποίες έχουν να χάσουν από αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ δύο λεπτά Είχα πει ένα λεπτό, λέει ο πρόεδρο, για την πρώτη ερώτηση. Ποιο θέλει να απαντήσει από του δημοσιογράφου, η κυρία Στάιν, σήκω στο χέρι, παρακαλώ. Μα πάντα. Ο, το χρήμα προσπαθεί να βρει μια διέξοδο, όπω και το νερό. Πάντα βρίσκει έναν δρόμο. Υπάρχουν πάντα τα συμφέροντα αυτά τα οποία ε, υπάρχουν σε όλες τις κυβερνήσεις και ίσως το γνωρίζετε καλύτερα από μένα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια χώρα να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά τη και γι' αυτό <clears throat> όταν δεν μπορεί να το πετύχει με άλλους τρόπους κανείς χρειάζεται να λειτουργήσει και σε ένα πιο διεθνές επίπεδο χρησιμοποιώντας εταιρείε γραμματοκιβατίου κτλ. Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες πώς θα μπορέσουν να δεσμευτούν όλες να σταματήσει μια τέτοια δραστηριότητα. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος θέλει να προσθέσει, κύριε Στρόντζικ. <coughs> θα ήθελα να σταθώ στο πρώτο ερώτημα για την έκταση του φαινομένου αυτού. Είδαμε στους φακέλους τα έγγραφα για τις Μπαχάμες. Βρήκαμε λιγότερα στοιχεία από ό,τι στην περίπτωση του Παναμά, αλλά βλέπουμε και πάλι ότι υπάρχουν χιλιάδες εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται. Είναι τη ίδια τάξη μεγέθους όπως για την περίπτωση του Παναμά. Εμείς δεν έχουμε απόλυτα αξιόπιστα στοιχεία, αλλά οι εμπειρογνώμονες λένε ότι αυτά τα οποία είδαμε τη Μόσακ Φονσέκα είναι ουσιαστικά ο τζίρο ενό έτου για αυτέ τι ε, εταιρείε. Μιλάμε για χιλιάδε επομένω εταιρείε. Αυτή είναι και η έκταση του φαινομένου. Λοιπόν, παρακαλώ. Θέλω να υπογραμμίσω ότι τα κύρια νομοθετικά βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν δεν εναπόκεινται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε αυτές τις χώρες που αναφέρθηκαν όπως είναι ο Παναμάς. Εκεί θα πρέπει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία των ε, εταιριών εκεί. Όταν λοιπόν δημιουργείται μια εταιρεία θα πρέπει να δημόσιε πληροφορίες ποιος έχει δημιουργήσει την εταιρεία και ποιοι είναι οι διευθυντές κτλ. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει μια πολιτική πίεση η οποία θα ασκηθεί στις χώρες αυτές. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο και ένα δεύτερο στοιχείο που είναι απαραίτητο είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. Ο ΩΣΑ έχει, όπως ξέρουμε όλοι, ξεκινήσει ένα εγχείρημα προς την κατεύθυνση αυτή <clears throat> για την ανταλλαγή πληροφοριών. Αλλά τα κύρια νομοθετικά βήματα τα οποία να γίνουν είναι εκτός της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς λοιπόν θα πρέπει να ασκήσουμε πρόταση, πίεση προς την κατεύθυνση αυτή. Ερχόμαστε τώρα στους ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες. Καταρχήν ο κ. Ρωσάτη, συντονιστή του ΕΛΚ, Και εγώ να ευχαριστήσω τους δημοσιογράφους που προσκαλέσαμε για τις τόσο διεξοδικές παρουσιάσεις και την ενδιαφέρουσα εικόνα Αυτή της παθολογικής θα έλεγα κατάστασης. Έχω δύο-τρεις ερωτήσεις, πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι τα βασικά κενά στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που έχετε εντοπίσει για την, στην οδηγία ειδικά για το ξέβλημα πλωμικού χρήματος και ίσως στις οδηγίες και τους κανονισμούς που αφορούν την ανταλλαγή φορολογικών δεδομένων και πληροφοριών που κατά την άποψη των προσκαλεσμένων μας θα μπορούσαν ε, να βελτιωθούν ή να αλλάξουν. Δεύτερη ερώτηση. Τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει σωστά την ευρωπαϊκή νομοθεσία και σε τι βαθμό Αυτές οι παθολογικές καταστάσεις που εντοπίστηκαν έχουν προξενηθεί από την πλημελή εφαρμογή, μεταφορά μάλλον της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και τέλος, γνωρίζουμε ότι το να δημιουργήσει κανείς ε, εταιρείε ε, φαντάσματα και να πάει σε φορολογικούς παραδείσους έχει το όφελος της ανωνυμίας και του κέρδους. Τι μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποτρέψουμε εδώ. Γιατί πρέπει να ασκήσουμε πολιτική πίεση, να διαπραγματευτούμε και ούτω καθεξής. Αλλά σε τι βαθμό από τη δική μας πλευρά μπορούμε να επιβάλλουμε υποχρέωση στους πολίτες και στις εταιρείε που έχουν έντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να καταγράφονται κάπου δραστηριότητε σε φορολογικού παραδείσους και ουσιατερίες. Ποιο θέλει να απαντήσει σε αυτό το δύσκολο ερώτημα. Πρέπει αυτό φυσικά να απαντηθεί και στο τέλος της εργασίας μας. Η κυρία Στάιν, να σας δώσω μια ένδειξη. Όπως είδαμε στη, στις περιπτώσεις του Πρωθυπουργού της ε, Ισλανδίας, έγιναν κάποιες ε, ενέργειες οι οποίες δεν είχαν να κάνουν με το νομικό πλαίσιο αλλά με την ηθική υποχρέωση των πολιτικών να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα. Επομένως, άμα με ρωτάτε τι πρέπει να αλλάξει σε νομικό επίπεδο, θα έπρεπε να υπάρχει ένα μητρό όπου να περιέχεται η πληροφορία για τους δικαιούχους και επίσης να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των χωρών, να συμμετέχουν όλε οι χώρε και άλλα και μέσα σε κάθε χώρα να εξασφαλίζεται ότι πράγματι λειτουργεί καλά αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο χρειάζονται περισσότερε προσπάθειε. Ευχαριστώ. Κύριε Τσίλμαν, δύο σημεία να αναφέρω εδώ. Έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ αυστηρούς ε, νόμου Αν αυτοί οι νόμοι εφαρμοζόντουσαν πλήρω θα είχαμε πολύ λιγότερα προβλήματα. Επομένω, ένα πρόβλημα είναι η εφαρμογή και η αστυνόμευση. Δεν βοηθάει να έχουμε ένα μητρό δικαιούχων όπως έχουμε στην Κύπρο όταν δεν είναι πραγματικοί δικαιούχοι. <clears throat> Αυτό δεν θα <clears throat> αλλάξει αν δεν υπάρξει σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας από τα κατημέρια. Και το δεύτερο είναι η προστασία των καταγγελόντων, των whistleblowers, σε τελική ανάλυση. <clears throat> είναι μονάχα αποκαλύψεις όπως αυτές των Panama Papers που αλλάζουν τα κατάσταση και αυτό γίνεται μονάχα εάν υπάρχει πραγματική προστασία για τους καταγγέλλοντες. Κυρία Κνούτ. Όπως είπε ο συνάδελφος, τα διαφανή μητρώα είναι ένα σημαντικό παράγοντας. Να υπάρχει διαφάνεια και περισσότερη συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών λόγω χάρη στην περίπτωση της Φινλανδίας αντί να επιτεθούν στα μέσα μαζική ενημέρωση, θα πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο από ό,τι κάνουν τώρα με άλλε αρχέ και να συνεχίσουν αυτέ τι έρευνε. Ευχαριστώ. Ακόμη 45 δευτερόλεπτα παρακαλώ για ερώτηση. Νταρίους. Αν έπρεπε να κάνετε μια blacklist, ένα μαύρο κατάλογο με χώρες που θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνα ως πρώτη προτεραιότητα, σε αυτή την υπόθεση, επειδή υπάρχουν υποψίε ότι είναι φορολογική παράδειση, τέλο πάντων ιδιαίτερα φιλικέ προ τι περιπτώσει και όσου προσπαθούν να κάνουν φοροδιαφυγή και φοροαπάτη. Τι, τι θα προτείνατε στην Επιτροπή αυτή, πρέπει να διοργανωθούμε κάπω. Και μάλλον θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε χώρε όπου αυτές οι πρακτικές είναι πολύ συνηθισμένες. Για να έχουμε και κάποιο σοβαρό αντίκτυπο. Τι θα προτείνατε. Μπορεί παρακαλώ κανείς ακόμη να δώσει μια σύντομη απάντηση. Παρακαλώ. Εντάξει, θα το συμπεριλάβουμε ως θέμα στις περαιτέρω συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτος ε, ο μιλητής του, των Σελστών, ε, Πέτερ Ζήμων. Ευχαριστώ. Πρώτη ερώτηση στον κύριο Στρότσικ. Αναφερθήκατε στις, ε, στα ταμιευτήρια των ομοσπόνδων κρατών είπατε ότι έχουν εμπλακεί τα Landesbank της Γερμανίας σε αυτά που λέει ο κύριος Ομπερμάερ αναφέρονται διάφορες συγκεκριμένε τέτοιες τράπεζες εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις τώρα γιατί είπατε στο παρελθόν και θα ήθελα να μου πείτε και ποιοι ήταν οι πελάτες γιατί αυτές οι τράπεζες, οι Landesbank ε, έχουν καθήκον να βοηθούν ορισμένους συγκεκριμένους πελάτες, για παράδειγμα, για να αναπτυχθεί η οικονομία του αντιστοίχου όμως του κράτους. Ξέρετε ποιες τέτοιες ε, τράπεζες μπορεί να έχουν εμπλακεί. Ο κύριος Τρότσικ, ναι, έχετε δίκιο. Από ό,τι ξέρουμε, δεν αφορά μόνο ορισμένες τέτοιες Landesbank, αλλά και άλλες τράπεζες. Αν συνεχίζουν να το κάνουν, δεν είμαι σε θέση να σας πω. Αλλά βρήκαμε περιπτώσεις όπου τέτοιες Landesbank ή άλλες τράπεζες που έχουν διασωθεί με δημόσιους πόρους πολύ πρόσφατα έχουν κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή όχι πριν από πέντε χρόνια αλλά νωρίτερα. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι παρόμοιος ε, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άλλες τράπεζες, ε, διάφορες θηγατρικές στο Λουξεμβούργο, την Ελβετία και στην περίπτωση της εταιρείας HSH Nordbank αφορά ακριβώς τους πελάτες ε, με πολλά περιουσιακά στοιχεία, τους πολύ πλούσιους πελάτες. Ορισμένες τράπεζες επίσης ε, εμπλέκονται ιδιαίτερα στον ναυτιλιακό τομέα. Και όπως θα ξέρετε η ναυτιλία έχει μεγάλη σχέση με αυτές τις υπεράκτες εταιρείε. Υπάρχουν πολλά στοιχεία στα έγγραφα του Παναμά για αυτά τα θέματα της ναυτιλίας από πλευρά ε, ποσοτικής ε, παίζουν μεγάλο ρόλο. Οι τράπεζες λοιπόν αυτέ λειτουργούν περίπου όπω όλες οι άλλες. Ευχαριστώ πολύ. Συμπλήρωμα, όχι. Πέτερ, θε να πει τίποτα άλλο. Δεύτερη ερώτηση. Προς τον κύριο Τσίλμαν. Για αυτά που είπε ότι στην ουσία πετάει ο ένα στον άλλο τον μπαλάκι της δέουσας επιμέλεια θα έπρεπε να γίνεται στον Παναμά, ε, στον Παναμά λένε έπρεπε να γίνεται στην Ελβετία, στην Ελβετία υπάρχει παρατηρά, παραθυράκι που τους επιτρέπει να μην την κάνουν. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε προδιαγραφές για παράδειγμα για την νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος. Ασχοληθήκατε με παραβάσεις που έχουν κάνει μεγάλες τέσσερις εταιρείε λογιστικού ελέγχου που έχουν υποχρεώσεις δέωσης επιμέλειας. Απάντηση, ναι, το αντιμετώπισα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που λένε ότι ένας δικηγόρος είναι υπεύθυνο για τη δέουσα επιμέλεια ακόμη και αν δεν υπογράφει. Αυτό εφαρμόζεται σε πολλές χώρες και στη Γερμανία, αλλά όχι στην Ελβετία. Γι' αυτό χρησιμοποιούν ε, Ελβετούς δικηγόρους και διαπιστώσαμε ότι το 2015, όχι για παλιότερες χρονιές, το 90% των εταιριών που ήταν ακόμη ενεργές και τις οποίες διαχειριζόταν η Mossack Fonseca χρησιμοποιούν το κόλπο με τους εικονικούς διευθυντές. Στη Γερμανία όμως δεν βρήκαμε κάτι τέτοιο. Στην Ελβετία ορισμένοι το κάνουν. Πολλοί μάλιστα στη Γενέβη. Και στην ουσία είναι μερικές δεκάδες ονόματα. Είναι λοιπόν περιορισμένοι αυτοί που ασχολούνται με αυτό το κλάδο στην Ελβετία, αλλά είναι πολύ επικερδής η δραστηριότητά τους. Παρακαλώ. Να προσθέσω και το εξή ακόμα άλλη μια περίπτωση στη Γερμανία. Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί, υπάρχει μια τράπεζα στο Αμβούργο που σε μια εταιρεία έχει ένα μερίδιο 25% και εδώ υπάρχει ο κανονισμός για το 25% συν 1. Δηλαδή είναι μια εταιρεία η οποία υπόκειται σε έλεγχο για αυτό το γεγονός για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό τον, ε, το, τους κανόνες έχει μια εταιρεία με την οποία συνεργάζεται και έτσι δεν φτάνει το 25% και δεν χρειάζεται να δεν είναι υπόχρεα ελέγχου. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται πολύ συχνά. Ευχαριστώ, Λεοπρόδος. Ο Πέτερ. Έχεις τρία δευτερόλεπτα ακόμα. Όχι. Η κυρία Ρου Όνεν έχει το λόγο από την ομάδα του ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους δημοσιογράφους που είναι εδώ παρόντες για το έργο το οποίο έχουν φέρει σε πέρας. Ελπίζω ότι η Ένωση των Ερευνητών Δημοσιογράφων, το ICIJ και η ετέτου θα συνεχίσουν το έργο του. Έχω ένα ερώτημα για τι ε, προκλήσει τη πρόσβαση σε πληροφορία και τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει την κατάσταση στα θέματα αυτά. Τα έγγραφα του Παναμά ήταν ένα, μια περίπτωση διαρροής χωρίς προηγούμενο για στοιχεία από εταιρείες offshore. Αλλά τα δεδομένα μόνο των Panama Papers δεν είναι επαρκή. Θα πρέπει να βρούμε και τα αντίστοιχα δεδομένα από διεθνείς τράπεζες δεδομένων και διεθνή μητρώα. Και το ερώτημα μου είναι, είχατε δυσκολίες για να αναζητήσετε τον τελικό κάτοχο και να πάρετε πληροφορίες για τα θέματα αυτά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει για να βελτιώσει τη διαφάνεια πληροφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες είναι θετικές σε ό,τι αφορά την πρακτική αυτή και θα πρέπει αυτές οι πρακτικές να μεταλαμπαδευτούν και αλλού. Στην Φιλανδία έχει γίνει μια ε, μεγάλη πίεση για να υπάρξει κατάργηση του συστήματος που επικρατούσε και να υπάρχει το σύστημα των εικονικών διευθυντών και στη Φιλανδία. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί το σύστημα της Φιλανδίας, αντίθετα θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες και ακόμα και οι οργανώσεις των επενδυτών συμφωνούν ότι αυτό είναι σωστό. Γνωρίζετε λοιπόν το ανοιχτό σύστημα, το διαφανές σύστημα για τους ε, ε, ιδιοκτήτες στη Φιλανδία. Ποιος θέλει να απαντήσει, η κυρία Κνούσου. πάρα πολύ σύντομα και στα φιλανδικά θα απαντήσω τώρα αν θέλετε. Τα μητρώα είναι ένα σημαντικό θέμα. Είναι ένα ζήτημα ανεξάρτητο αυτό καθεαυτό. Υπάρχουν τώρα προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται στη Φιλανδία για να επιτραπεί οι Φιλανδοί δικαιούχοι να αποκρύπτουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ελπίζω ότι αυτή η νομοθεσία δεν θα ευδοκιμήσει, δεν θα περάσει στο Κοινοβούλιο στη Φιλανδία. Τα μητρώα του Παναμά δεν είναι ανοιχτά. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούν πάρα πολύ πάρα πολλές στα μητρώα του Παναμά γιατί δεν υπάρχει τρόπος με διαφάνεια να καταλάβει κανείς ποιος είναι ο πραγματικός κάτοχος. Αυτό συμβαίνει σε όλου του φορολογικού παραδείσου. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα μόνο όταν υπάρχει διαρροή εγγράφων. Αλλιώ δεν ξέρουμε τι ακριβώ γίνεται. Θέλει να απαντήσει κανεί από του δημοσιογράφου, ο κύριο Ζήλμαν. Θα μα βοηθούσε εάν ε, ήταν δημόσιο το Μητρό για τους ε, δικαιούχους ε, στον Παναμά ή στα Virgin Islands. Αυτό θα δυσχαίραινε τις τράπεζες και τους ενδιάμεσους που προσπαθούν να κρύψουν τους ε, πελάτες τους. Εκτός αν δεν υπάρχει λόγος να τους κρύψουν. Το ερώτημα όμως είναι εάν είναι ανοιχτό το μητρό μήπως θα χρησιμοποιούνται περισσότερο άτομα, βιτρίνα, αχυράνθρωποι περισσότερο. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει διαφάνεια λοιπόν αλλά μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχει και σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας. Πρέπει παράλληλα να λειτουργούν αυτά. Έχετε κι άλλη μία ερώτηση, έχετε άλλο ένα λεπτό. Πρόεδρε. Υπάρχουν ένα σωρό δεδομένα που έχουν διαρρεύσει και δείχνουν τι σημασία έχουν οι καταγγέλλοντες πληροφοριοδότες. Έχετε καμιά ιδέα για το τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους προστατεύσει τους whistleblowers. Και άλλη μία ερώτηση. Με τόσες διαρροές τελευταία, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μια σχετική κόπωση ο κόσμος και το κοινό να πάψει να ενδιαφέρεται για αυτού του είδους της αποκαλύψης. Θα μπορούσε να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να παραμείνει μεταξύ των καυτών ζητημάτων της επικυρότητας ε, το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ε, ποιος μπορεί να απαντήσει σε λίγα δευτερόλεπτα. Στάιν. Το Λουξεμβούργο είναι ιδρυτικό κράτος μέλος ε, της Ένωσης και δικάζονται δύο δημοσιογράφοι για τα LuxLeaks. Δεν είναι δυνατόν ε, να θεωρείται μικρότερο το δημόσιο συμφέρον από την προστασία κάποιων ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτές οι υποθέσεις καταδεικνύουν ότι οπωσδήποτε πρέπει οι whistleblower να προστατεύονται περισσότερο. Συμφωνώ, λέει ο Πρόεδρο. Επόμενο στον ομιλητή, ο συνάδελφο Μίχελ Τόιρερ από την Άλντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, ω συντονιστή τη Άλντε, θέλω να συγχαρώ του δημοσιογράφου και να του ευχαριστήσω για την εργασία του. Πρέπει οπωσδήποτε οι whistleblower να προστατεύονται καλύτερα. Αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο. Είναι κρίμα που δεν μας ακούει ο κύριος Όμπερ Μάιερ Ελπίζω όμως να ξανασυζητήσουμε αργότερα μαζί του. Ερώτηση προς την κυρία Στάιν και τον κύριο Στρότσικ. Αναφέρατε ότι αυτή η ενδιάμεση, για παράδειγμα στο Λουξεμβούργο, αλλά και στη Γερμανία και αλλού, δημιουργούν ε, διάφορες τέτοιες εταιρείε γράμματο κυβότιο για τους πελάτες τους. Θεωρείτε ότι ελέγχουν επαρκώς οι τράπεζες. Δηλαδή, βρήκατε ενδείξεις για παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Επίσης κύριε Στρότσικ είπατε ότι πολύ συχνά διαπιστώσατε ότι οι εργαζόμενοι στη Μόσακ ε, Φονσέκα είχαν και προσωπικές σχέσεις με διάφορους ενδιάμεσους. Ε, είδατε μήπως ένας γιος Φονσέκα εργαζόταν σε μια γερμανική τράπεζα, το διαπιστώσατε αυτό. Και μπορέσετε να μιλήσετε με τον Γιούργεν Μόσακ. Θέσατε τα θέματα αυτά στον κύριο Γιούργεν Μόσακ. Ευχαριστώ. Κύριε Στρότσικ, σε εσά απευθύνθηκε η ερώτηση. Βεβαίω, σε μένα. Ναι. Δεν μιλήσαμε με τον Γιούργεν Μόσακ. Μόνο γραπτό ανταλλάξαμε πληροφορίε. Είπαμε ότι ένα μέλος της οικογένειας Φονσέκα που είναι το δεύτερο μέλος ε, Μόσακ Φονσέκα. Δεν νομίζω πως ήταν γιος, ήταν ανιψιός του ιδιοκτήτη της Μόσακ Φονσέκα. Ε, είχε κάνει μία μαθητεία σε μία ελβετική θηγατρική, σε ένα ελβετικό υποκατάστημα γερμανικής τράπεζας. Αλλά δεν είναι σαφές. Δεν ήταν απόλυτα σαφέ αν συνέβη κάτι τέτοιο. Υπήρξε αμφισβήτηση. Κάτι άλλο να πω, μιλήσω λίγο ευρύτερα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτού του τύπου δραστηριότητε και από πλευρά τραπεζών και από πλευρά ενδιαμέσων και δικηγόρων κτλ. Και, και από πλευρά της Μοσάκ Φονσέκα Όλα αυτά γίνονται ε, σε μεγάλο βαθμό από Γερμανούς ή από ανθρώπους που καταλαβαίνουν γερμανικά υπήρχε για μεγάλο βαθμό η τράπεζα Δρέσδη Λατινική Αμερική, Δρέσνα Λατάιν Αμέρικα και πολλοί Γερμανοί εργαζόμενοι στον τραπεζικό τομέα και κυρίως με έδρα στο Στρασβούργο και διάφορα ταμιευτήρια που άρχισαν να έχουν δραστηριότητα και στη Λατινική Αμερική και από εκεί ήρθα σε επαφή με τη Μοσάκ Φονσέκα και διάφοροι από αυτή την ε, τράπεζα της Δρέσδης πήγανε και στην τράπεζα Μπέρναρ κτλ. Όλοι αυτοί, ξέρετε, πολλές φορές ε, δούλευαν ε, ο ένας στον έναν όροφο, ο άλλος στον άλλο, έκαναν μαζί διακοπές οικογένειές τους. Δηλαδή δεν είχαν μόνο επαγγελματικές σχέσεις, δεν συναντιόνταν μόνο σε συνέδρια. Αλλά γενικότερα όλοι όσοι προέρχονταν από αυτή την τράπεζα στην Δρέσδη έπαιξαν μεγάλο ρόλο ούτω ώστε ε, το γραφείο Mossack Fonseca να έχει τόσε σχέσει με τη Γερμανία και με την Ελβετία. Συμπλήρωση, λέει ο πρόεδρο, όχι, δεν υπάρχει. Μίχαλ Τόερα, έχετε ακόμη ένα λεπτό 20 δευτερόλεπτα. Ένα ακόμα ερώτημα, ένα πρόσθετο ερώτημα. Κύριε Στρότσεξ, σε ό,τι αφορά την εποπτεία των τραπεζών, είπατε ότι είναι σημαντικό ο ρόλο των τραπεζών και η κυρία Κνούστο ανέφερε αυτό ότι υπήρχε μια διαδικασία κυκλική ε, ε, κυκλικών συναλλαγών, καρουσέλ. Υπάρχουν τώρα στοιχεία που να δείχνουν ότι έχει αστοχήσει η τραπεζική εποπτεία ή υπάρχει ένα πρόβλημα νομοθετικό. Ευχαριστώ ποιος από τους δημοσιογράφους θα ήθελε να δώσει μια απάντηση, η οποία φυσικά είναι μια ερώτηση πρέπει να, να την απευθύνουμε περισσότερο στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως οι αρχές αυτές πολλές φορές έκαναν σαν να μην ήταν καθήκον τους να εξασφαλίσουν τα θέματα αυτά και εμείς ως δημοσιογράφοι δεν βρήκαμε να έχουν υπάρξει, να υπάρξει διαφάνεια στο βαθμό που θέλαμε. Ο κύριος Στρότσικ θα μπορούσε ναι. Ναι. Με την Buffen μπορώ να, για την Buffen μπορώ να αναφερθώ την υποπτική υπηρεσία για τις γερμανικές εταιρείες. Μπορεί πάντα να εξασφαλίσει τον έλεγχο του workflow στις ε, τράπεζες αν υπάρχει η πρέπουσα επιμέλεια για τα θέματα αυτά, αν έχει γίνει ο έλεγχος ο οποίος είναι απαραίτητος και μπορεί με τον τρόπο αυτό να δει αν οι πληροφορίες που δίδονται στην εποπτική αρχή είναι σωστές ή όχι. Ο ρόλος της Μπάφεν όμως δεν είναι επαρκής για να μπορέσει να ελέγξει αυτά τα πράγματα, ελέγχει τη λειτουργικότητα των συστημάτων στι τράπεζε. Αυτό για μένα δεν είναι επαρκέ, αλλά σίγουρα εμεί θέλουμε περισσότερε δυνατότητε για αυτήν την Μπάφεν στην Γερμανία. Ακολουθεί ο, ο κύριο Κούλογλου από την ΚΟΕ. Παρακαλώ. Well, uh, I think it's very important that... Νομίζω είναι πολύ σημαντικό ό,τι μας είπαν και εξήγησαν οι δημοσιογράφοι εδώ. Είναι σημαντικό να εντοπίσουμε το ρόλο των καταγγελόντων και να μπορέσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να τους προστατεύσουμε. Πρέπει σε ανθρώπους όπως αυτοί που μας ε, εντόπισαν την περίπτωση LuxLeaks να μην καταδικαστούν, να μην διωχθούν, να μην φτάσουν στα δικαστήρια. Ο Σνόντεν άνοιξε τον δρόμο. Ο Άσερ άνοιξε το δρόμο για, την, ε, για τις καταγγελίες και την ε, παρόχεια πληροφοριών στη σύγχρονη περίοδο τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζετε και ήθελα να ρωτήσω όλους τους δημοσιογράφους Εδώ τα τελευταία χρόνια θα ξέρατε ότι ψηφίσαμε για την προστασία των, ε, της μυστικότητας της επιχειρήσης, στο απόρριτο της επιχειρήσης. Ήθελα να σας ρωτήσω εάν έχετε προτάσεις για την προστασία του δικαιώματος των δημοσιογράφων να ερευνούν τέτοιες περιπτώσεις και υποθέσεις. Έχετε ακριβείς ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε. να ψηφίσουμε υπέρ της διαφάνειας, της διευκόλυνσης του έργου σας. Αλλά με ποιες ιδέες για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Ποιος θέλει Maybe one, element. Ίσως ένα στοιχείο που θα μπορούσε να προσθεθεί σε αυτή τη συζήτηση είναι η σημαντική χρήση της ε, κρυπτογράφησης η κρυπτογράφηση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας ήταν μια από τις προτεραιότητες. Οι αρχές θα μπορούσαν να έχουν λοιπόν σε κρυπτογραφημένα δεδομένα πρόσβαση τα λεγόμενα encrypted, αλλά και εμείς πολλές φορές με κώδικα επικοινωνούμε μεταξύ μας, με encryption όπως λέγεται, ε, οι ερευνητές δημοσιογράφοι που συνεργαζόμαστε. Δεν είναι ε, μυστικό αυτό, ξέρουμε ότι πολλοί το κάνουν αυτό για να μην αφήνουν ίχνη πίσω τους, οπότε οι δημοσιογράφοι αν θέλουν για ευαίσθητα ζητήματα να ε, συζητήσουν μυστικά χωρίς να τους εντοπίσουν τρίτη, η ε, κωδικογράφηση αυτή, η κρυπτογράφηση είναι ένας πολύ καλός τρόπος. Ευχαριστώ. Θέλετε να θέσετε συμπληρωματικό ερώτημα. Ναι, να ρωτήσω τον κύριο Κλέριξ. Είπε ότι σε κάθε έρευνα η κλασική απάντηση ήταν αυτό που κάνουμε είναι στα πλαίσια του νόμου. Ήθελα να μου πείτε εάν Πιστεύετε ότι υπάρχουν νόμοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν ώστε όλο το σύστημα να γίνει πιο διαφανές και να διευκολυνθεί και η δικιά σα δουλειά. Ευχαριστώ κύριε Κλέριξ. Όπως είπα προηγουμένως, νομίζω ότι η κύρια νομοθεσία που πρέπει να αλλάξει είναι αυτή που ισχύει στους φορολογικούς παραδείσους, δηλαδή στις χώρες όπου η νομοθεσία εξασφαλίζει τη δυνατότητα ανωνυμίας. Εκεί είναι τα κύρια βήματα τα οποία θα πρέπει να, να γίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο εξάλλου όλα τα κράτη-μέλη να έχουν καλές εγγυήσεις για την προστασία των πηγών των δημοσιογράφων, ώστε έτσι να διευκολυνθεί και το έργο των δημοσιογράφων. Το Βέλγιο είναι καλό παράδειγμα από αυτή την άποψη. Σε ό,τι αφορά την προστασία των ε, καταγγελόντων, το whistleblower, υπάρχει το θέμα της προστασίας από δικαστική δίωξη στη συνέχεια και επίσης πρέπει να σκεφτούμε και το μέλλον της ζωής σας. Φανταστείτε ότι έχετε αποκαλύψει πληροφορίες από μια εταιρεία όπου εργαζόσατε και την επόμενη εβδομάδα σας έχουν απολύσει. Θα πρέπει να βρείτε μια νέα δουλειά. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ανάγκη της προστασίας του μέλλοντος των καταγγελών να υπάρξει και ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος γύρος ομιλητών, Σβέν Γκίγκολτ πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. θεωρούμε ότι αυτή η Εξεταστική Επιτροπή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να καθαρίσουμε την κόπρο του Αυγίου της ε, μυστικότητας ε, σε αυτές τις συναλλαγές. Αλλά δεν προστατεύονται επαρκώς οι whistleblower και προς τον Jean-Claude Juncker απευθυνόμενος. Θέλω να πω ότι δεν θέλουμε μια νέα διαβούλευση για την προστασία τους. Θέλουμε νομοθετική πρόταση και τη θέλουμε εδώ και τώρα. Τώρα στις 12 σε μια συνέντευξη τύπου θα παρουσιάσουμε το λογισμικό EU Leaks που επιτρέπει σε όποιον whistleblower θέλει να ε, αποστείλει μυστικά στοιχεία για οποιαδήποτε ενδεχόμενα οικονομικών εγκλημάτων στα κράτη-μέλη, τον ιδιωτικό τομέα, την Ένωση και επίση για περιπτώσεις, για παράδειγμα, κακοδίκησης ή παράβαση γενικότερα του ενωσιακού νόμου. Θέλω να ρωτήσω του ε, δημοσιογράφους. Είχατε καμία γνώση τέτοιων περιπτώσεων. Μπορείτε να μας πείτε εάν είδατε τέτοιες ε, περιπτώσεις κακοδίκησης ή παράβασης του νόμου. Ευχαριστώ. Ποιος θα ξεκινήσει, λέει Πρόεδρος. Μπορώ να μιλήσω μόνο για αυτά τα οποία ερεύνησα. Είδαμε παρεμβιάσει του νόμου στην ε, Κύπρο, όπου δεν αναφέρονταν οι πραγματικοί δικαιούχοι και ε, ήρθαμε σε επαφή με τις ρωσικές τράπεζες στην Κύπρο και μας είπαν όλες αυτές τις βλακίες. Δεν μας έδωσαν ουσιαστικές απαντήσεις. Άρα μπορούμε να διαρμηνήσουμε περδέρω αυτές τις υποθέσεις. και από ό,τι θυμάμαι το 2008-2009 ήταν έγκλημα να μην αναφέρει το πραγματικός δικαιούχος και σε πολύ λίγες περιπτώσεις υπάρχουν κυρώσεις εάν κάποιος αναφέρει ψευδή πραγματικό δικαιούχο. Τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να τιμωρούνται και να αναφερθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει να συμπληρώσει. Η κυρία Κνούς. Στις περιπτώσεις ξεπλήματος της Μέτσο, το μόνο που έγινε ήταν να απολύθηκε ο διευθυντής. Η αστυνομία όμως δεν ερευνά την υπόθεση, όπως έχω πει. Περίεργο, θα φανταζόταν κανείς ότι ότι αυτό είχε να κάνει με τη Ρωσία επειδή είναι Ρώσος και ότι αφορά πολλές διαφορετικές δικαιοδοσίες και νομοθεσίες. Το βρίσκω παράξενο να συμβαίνει στην Ευρώπη και κανείς να μην ερευνά. Παραβιάσεις του νόμου, εάν μιλάμε για την προστασία των πηγών λόγου χάρη, όπως σας είπα στην Φιλανδία, ως τώρα ήταν πάρα πολύ καλό το ιστορικό μας. έξι ε, εξαετή κάθερξη μπορεί να έχει κανείς ε, για την απόκρυψη στοιχείων, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στα διοικητικά δικαστήρια και θα δούμε αν αλλάξει το σύστημα προστασίας των πηγών στη Φιλανδία. Άλλος να πει κάτι? Απλώς να πω ότι σε μια συνέντευξη που έκανα ε, με την Europro, την, ε, το σώμα της Ευρώπης για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, ε, όταν ερευνούσαμε το θέμα του Panama Papers, είπαν ότι η Europol δεν κάνει καμία έρευνα για τις χρηματοοικονομικές αυτές απάτες. Έχουν δύο offshore και τις ξέρουν εδώ και καιρό. Καλέστε τους εδώ σε αυτήν την Επιτροπή σα όχι μόνο για την περίπτωση της Μόσακ Φονσέκα του Λουξεμβούργου, αλλά γενικότερα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, για τους φοροφυγάντες, για ότι θα μπορούσαν να σα πούνε ποιοι είναι οι νόμοι που παραβιάζονται. Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να γράψουν τόσο εύκολα ένα άρθρο για κάποιον που παρανομεί επώνυμα, μπορούμε να γράψουμε για αυτά που βλέπουμε, μπορούμε να γράψουμε για αποδεικτικά στοιχεία που μπορεί να έχουμε εφόσον έχουμε έγγραφα στα χέρια μα. Όμω είναι βασικά ρόλο των εισαγγελέων και των ερωτητών δικαστών να εντοπίσουν τα έγγραφα και να θέσουν το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων για το πού ακριβώ έγινε η παραβίαση του νόμου. Η Europol λοιπόν θα μπορούσε να συνεισφέρει στην έρευνά σα. Σα ευχαριστώ πολύ. Λίγα δευτερόλεπτα έχουμε. Ο Ντέβιτ Κόμπον γιατί το EFTD έχει το λόγο τώρα. Να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι κάτι που είναι γνωστό σε πολλούς από εμά. δίποτε βρίσκεται στον επιχειρηματικό κόσμο τα γνώριζε αυτά. Γι' αυτό θέλω να θέσω το εξή ερώτημα στους δημοσιογράφους. Είναι πρόβλημα αυτό το ξέπλυμα χρημάτων θα ήθελα φυσικά να αποκαλυφθεί από τους καταγγέλλοντες, αλλά μπορεί η καταγγελία να είναι θεμητή, αλλά αν οποιοδήποτε αποφασίσει σε μια τράπεζα να δίνει εμπιστευτικές πληροφορίες δεξιά και αριστερά, όλο το τραπεζικό οικοδόμημα καταραίει. Πρέπει να υπάρχει και κάποιο στοιχείο για την ε, υπευθυνότητα και των δημοσιογράφων και των καταγγελόντων. Είναι πάρα πολλοί λοιπόν οι οποίοι μπορούν να βρουν μια δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από μια καταγγελία. Θα ήθελα να ξέρω όμω πώ θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα τη προστασία των καταγγελόντων. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει και προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Ποιος θέλει να απαντήσει, κυρία Στάιν, πρώτα. Εγώ δεν θέλω να νομιμοποιήσω την ε, αποκάλυψη τραπεζικών μυστικών. Αλλά αν δείτε τι έγινε στην περίπτωση του Λουξεμβούργου. Μόλις αναποκαλύφθηκαν τα Lux Leaks, δύο δημοσιογράφοι βρέθηκαν ενώπιον των δικαστήριων. Και αυτό ήταν αντίθετο με το ένομο συμφέρον όλων των πολιτών, το ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου. Γιατί αυτοί αποκαλύπτουν φορολογικές παραβιάσεις οι οποίες θίγουν όλους τους Ευρωπαίους. Επομένως εδώ φαίνεται ότι ήταν λανθασμένη, ότι ήταν στρεβλή αυτή η διαδικασία που οδηγεί τους καταγγέλλοντες στο δικαστήριο. Ευχαριστώ. Το βασικό σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να τονίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Πρέπει να υπάρξει επικράτηση του δημοσίου συμφέροντο. Και αυτό το έχει τονίσει το ΕΔΑ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεν είναι φυσικά ότι οποιοδήποτε μυστικό μπορεί να γίνει δημόσιο, αλλά όταν εμπλέκεται το δημόσιο συμφέρον, όπω ήταν ακριβώ η περίπτωση για τα έγγραφα του Παναμά και τα LuxLeaks, τότε πρέπει να υπερέχει το δημόσιο συμφέρον και να υπάρχουν εξαιρέσει σε αυτέ τι περιπτώσει. Στρότσικ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, όχι. Έχετε ένα πρόσθετο ερώτημα να θέσετε. Παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο μιλητής. Συγγνώμη. Ήταν ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό σαν ένα πρόσχημα για να διευρύνει την επιρροή της σε όλο τον κόσμο. Μα βέβαια το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο μιλητής. Εμείς θα φύγουμε βέβαια, αλλά το πρόβλημα είναι ότι βάζουν τη μύτη τους, χώνουν τη μύτη τους παντού. μήπως θα μπορούσαν τα κάτι μελη να το αντιμετωπίσουν στο εσωτερικό τους καθεμία και όχι να αφήνουν ε, τις, ευρωπαϊκέ ευρωπαϊκές αρχές να απλώνουν τα πλοκάμια τους δεξιά και αριστερά. Μα έχουμε και κάποια απικία, έχουμε κάποιες απικίες της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου που παίζουν ρόλο σε όλα αυτά. Ο κύριος Τσίλμαν. Νομίζω είναι η πέμπτη αποκάλυψη που είχαμε για εταιρείε ε, offshore. Είχαμε αποκάλυψη για το Λουξεμβούργο, για την Ελβετία, για την Κίνα, για τον Παναμά. όλο μας λένε ότι ο καθένα πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του και να μην επεμβαίνει σε άλλε περιπτώσει, Αλλά κάθε περίπτωση καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρξει μια γενικότερη ρύθμιση, ακόμα και αν είναι κανεί εναντίον. Εμεί όμω δεν μπορούμε αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε την, ε, τις offshore, είναι ουσιαστικά το Wild West, δηλαδή κάνει ο καθένας ό,τι, ό,τι του κατεβαίνει εκεί πέρα. Δεν υπάρχει καμία α, μορφή ελέγχου. Έχουμε παγκόσμια φαινόμενα όπως είναι η, η τρομοκρατία, τα αδικήματα παιδοφιλίας παγκοσχάρη αντίον το παιδιών ή το υπερική πορνογραφία. Όλα αυτά είναι εγκλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν γενικότερα. Ευχαριστώ. Η το παιδική πορνογραφια ολα αυτα Μπάρμπαρα Κάπελ κυρια Μπάρβαρα καπελ απο την ε, ΕΔΕ. Κύριε Κόμπερν, 30 δευτερόλεπτα έχετε ακόμα. Όχι, δεν θέλετε. Κάπελ. Κύριε Κνούς, αυτό που είπατε για τις διαρροές, το δημόσιο συμφέρον, όπως είπε και η Τζούλια και ο Χριστόφ, αυτή είναι η βασική έννοια. Γι' αυτό οι δημοσιογράφοι όταν κάνουν έρευνες πρέπει να εξετάζουν το περιεχόμενο των διαρροών δεν ε, ανεβάζεις απλώς το, όλες τις διαρροές ε, στο ίντερνετ. Ε, τι θα κάνετε για παράδειγμα λοιπόν με αυτό το νέο site, εάν κάποιοι βάλουν στοιχεία, θα πρέπει κάποιος να τα μελετήσει, να τα αξιοποιήσει για να δει εάν υπάρχει δημόσιο συμφέρον. Το θέμα λοιπόν είναι να δούμε αν υπάρχει δημόσιο συμφέρον, όχι απλώς να πετάμε κάτι στο ίντερνετ. Ευχαριστώ κυρία Κάπελα από το ENF, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, και αυτού του ομίλου δημοσιογράφων, ICIG. Καταφέρατε να αποκαλύψετε ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο και μελετήσατε 11,5 εκατομμύρια έγγραφα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει καθαυμασμός για την εργασία σας. Και το σημαντικότερο είναι ότι καταφέρατε να μπει στο ενδιαφέρον στη κοινή, της κοινής γνώμης, ούτως ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Διότι, όπως ξέρετε, οι προϋπολογισμοί της Ένωσης και των κρατών μελών χάνουν 70 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο από φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. όλα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό υπάρχουν διάφορα πακέτα για την αντιμετώπιση αυτό το φαινομένων και είναι πολύ σημαντική η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει περισσότερη αποτελεσματικότητα και περισσότερη δικαιοσύνη στα φορολογικά συστήματα. Τα μέτρα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη διεθνή προσπάθεια. Υπάρχουν ε, τα σχέδια δράσης BEPS των 15 σημείων και στη συνάντηση κορυφή στη Χανζού υπόθηκε ότι πρέπει ο ΩΣΑ να καταρτήσει ένα κατάλογο όλων των φορολογικών παραδείσων. Ξέρουμε ότι οι τρεις μεγαλύτεροι φορολογικοί παράδοσοι που είναι η Ελβετία, οι Ηνωμένε Πολιτείε και το Ηνωμένο Βασίλειο και τα εξαρτώμενα εδάφη του πρέπει να σταματήσουν να δρουν όπως δρουν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας κατάλογος και αυτό είναι το ερώτημά μου Θέλετε να επιτύχουμε να εφαρμόζεται ο νόμος και σε αυτά τα κράτη που προανέφερα. Επίσης, είπατε ότι πρέπει να υπάρχει και ένας ε, κώδικας διοντολογίας για τις τράπεζες και τους ε, φορολογικούς συμβούλους. Αυτό το αναφέρει και το πόρισμα της Επιτροπής Τάξε. Τι γνώμη έχετε από αυτού. Επαρκούν όλα αυτά, επαρκεί ένας κώδικας δεντολογίας ή θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερα μέτρα εφαρμογής του νόμου, πολύ περισσότερα από αυτά που έχουμε ήδη. Κυρία Κάπελ, αντί για ένα λεπτό μιλήσατε δύο λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ποιος θα απαντήσει, ο κύριος Τρότσικ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχει νομοθεσία, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι αφορούν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την πρέπουσα επιμέλεια. Και συγχρόνως έχουμε γνωρίζουμε τις ιστορίες που έχουν γίνει με την Ελβετία και το Λουξεμβούργο για την αποκάλυψη τεθών κτλ. Πρέπει να δούμε λοιπόν όταν θεσπίσουμε κάποιο κώδικα τι θα προκύψει. Αν είναι καλά λειτουργών θα μπορέσει να μας επιτρέψει να αποκαλύψουμε κάποια πράγματα. Αν όχι, θα δούμε ότι αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ξέρουμε ότι πολλές μεγάλες τράπεζες έχουν παίξει ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και θα πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία που γίνεται μέσω αυτών. Ποιο θέλει να προσθέσει κάτι, Τσίλμαν. Ναι. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν μαύροι κατάλογοι και χώρες όπως η Ελβετία έχουν κάνει μεγάλες πρόοδους στα θέματα αυτά και έχουν λειτουργήσει αυτά, αλλά έχουμε πάρα πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τους ε, δικηγόρους. Όλοι οι διεθνείς ε, ενδιάμεση θα πρέπει να υπόκειται σε πιο έντονο έλεγχο. Έχω λοιπόν τι εξή προτάσεις. Βοηθάει το να φτιάμε μαύρους καταλόγους, αλλά ό,τι χρειάζεται και αυτό φάνηκε και από την ε, περίπτωση που είδαμε της Κύπρου και της Ελβετίας να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα παραθυράκια. Υπάρχουν πολλές τράπεζες επίσης που έχουν διασωθεί και οι οποίες έχουν εμπλακεί σε αυτή την ε, περίπτωση δεν μπορούμε αναδρομικά να καλύψουμε τα πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν, θα πρέπει τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Ναι, δυστυχώ η πολιτική βρίσκεται σε μια υστέρηση πολλέ φορέ από αυτά τα φαινόμενα. Ο κύριο Ρούντρικ Νίτερμαερ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου αυτού του δημοσιογράφου που έχουν έλθει ενώπιόν μα και μα βοηθούν να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα όχι μόνο για μερικούς αλλά για όλους. Έρχομαι στην εκκίνηση της συζήτησης. Ελπίζω ότι με την εργασία της Επιτροπής μας θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πολύ καλύτερα τι έχει συμβεί. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ποια είναι η ουσία και όχι μονάχα τα επιφαινόμενα. Ξέρουμε ότι γίνονται πολλά πράγματα τα οποία γίνονται κάτω από τη μύτη μας όπως είπαμε πολλοί δημοσιογράφοι. Δεν είναι επαρκές να πούμε ότι κάποιοι ενδιαφέροντες άνθρωποι έχουν πολλά χρήματα σε κάποια εξωτικά μέρη του κόσμου. Πρέπει να καταλάβουμε τι υπάρχει πίσω από όλα αυτά. Ξεκινώ λοιπόν με δύο απλές ερωτήσεις που θέλω να θέσω. Πρώτα απ' όλα, μετά από τις αποκαλύψεις των LuxLeaks και των εγγράφων του Παναμά, στην περίπτωση του LuxLeaks τα πράγματα ήταν απλά Είχαμε εταιρείε οι οποίε με επιθετικό τρόπο προσπαθούν να εξασφαλίσουν την φόρο αποφυγή και αυτό μπορούσε να γίνει λόγω των παραθυρακίων που ήταν στην ε, νομοθεσία τη φορολογία. Ενώ είναι πιο πολύπλοκο το θέμα ε, των εγγράφων του Παναμά που αποκαλύπτουν διαφθορά, έκπληση χρημάτων και δραστηριότητε που είναι στο όριο του νόμιου είναι και παράνομε. Το πρώτο ερώτημά μου είναι λοιπόν αν Θεωρείτε ότι είναι πιο πολύπλοκη η περίπτωση των Panama Papers και δεύτερο ερώτημα. Κατά τη δική σας κρίση πιστεύετε ότι ο κύριος στόχος αυτών των δραστηριοτήτων που έχετε αποκαλύψει στην έκθεσή σας είναι κυρίως παράνομες ε, δραστηριότητες οι οποίες συγκαλύπτονται ή απλώς η φοροδιαφυγή για τους πλούσιους ιδιοκτήτες εταιριών ή βλέπετε κυρίως νόμιμες δραστηριότητες αλλά ιδιαίτερα με σε ηθικό επίπεδο δραστηριότητες που επιτρέπουν σε κάποιους να βγάλουν τα κέρδη τους από ε, περιοχές όπου υπάρχει ε, πραγματική φορολογική εξουσία σε άλλες ε, περιοχές. Κύριε Στάιν. Μα είναι εντελώ διαφορετικές δραστηριότητες. Νομίζω ότι κατέστη σαφές. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν σε κάθε χώρα διάφοροι μεσαίου εισοδήματος που θέλουν να πληρώσουν λιγότερο φόρο. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις ε, κρύβονται και εγκληματικές δραστηριότητες. Πόσο περίπλοκα είναι όλα αυτά τα θέματα για μας. Τα έγγραφα του Παναμά δεν ήταν και τόσο πιο περίπλοκα, γιατί ήταν πλούσιο το υλικό. Άρα διευκόλυνε τη δουλειά μας. Πλουσιότερο και από πλευράς περιεχομένου σε σχέση με το LuxLeaks. Αλλά, όπως σωστά είπατε κι εσείς, στην περίπτωση του Λουξεμβούργου ήταν ε, τα διάφορα παραθυράκια για την ε, αποφυγή του φόρου, ενώ στην περίπτωση του Παναμά ήταν διαφορετική η περίπτωση. Για παράδειγμα, διάφοροι πολιτικοί οι οποίοι δεν ήταν πια θέσει εξουσία προθώσαν να κρύψουν ε, κάποια εισοδήματα. Άρα είναι περισσότερο ε, λόγοι ιδεοντολογία, ηθική. Γι' αυτό είναι μεγαλύτερη πρόκληση για να δούμε τι μπορούμε να αναφέρουμε, από ποια οπτική γωνία πρέπει να τονίσουμε αυτό το θέμα για να σταματήσουν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Κλέρεξ. Συμφωνώ με την ε, Τζούλια. Η περίπτωση LuxLeaks ήταν πολύ πιο περίπλοκη. Δεν ξέρω αν κανεί μπήκε στην, ε, στον κόπο να διαβάσει τι δικαστικέ αποφάσει ε, και τι δικαστικέ συμφωνίε, αλλά πραγματικά ήταν πυρηνική φυσική. Ήταν πάρα πολύ κεφαλική και λαβυρινθώδηση επεξεργασία όλου αυτού του συστήματο. Είναι διαφορετικέ αυτέ λοιπόν οι φορολογικέ συμφωνίε, οι μυστικέ. Το Panama Papers έχει να κάνει με την εξή απλή αρχή θέλω να βγω εκτός των προβολέων. Δεν θέλω να συνδέομαι με αυτό το μεγάλο τραπεζικό λογαριασμό, ε, ούτε τα χρήματά μου να φαίνεται από πού προήλθαν. Θέλω μια ανώνυμη εταιρεία και να βγω εκτός. Αυτό έγινε επειδή το επέτρεψαν 21 δικαιοδοσίες ουσιαστικά. Είναι σαφές, είναι ξεκάθαρο και ευνόητο. Τώρα, ποιοι ήταν οι σκοποί, παράνομοι και νομότυποι. Να αναφέρω κάτι που είπε ο κύριος Δελαπιέρ σε μια συνέντευξη από την Βελγική Αρχή για, κατά του ξαπλήματος βρώμικου χρήματος, ότι σε όλη μου τη ζωή δεν είδα κανέναν να ε, φτιάχνει ε, εταιρεία offshore για περισσότερη διαφάνεια. Αυτό είναι το ζουμί. Εάν ήθελε κανείς να τη χρησιμοποιήσει για νόμιμους σκοπούς, ε, τι θα την έκανε άλλο από το να κρύψει κάτι. Ε, τι λόγους έχει κάποιος να κρύψει κάτι. Από τον ε, συνεταίρο του θα μπορούσε να θέλει να κρύψει κάτι κανείς, γιατί δεν συμφωνεί με τη στρατηγική του, αλλά αυτό δεν είναι παρανομία. Ε, μπορεί κανείς να θέλει να κρύψει περιουσιακά στοιχεία σε ένα διαζύγιο, για τη μελλοντική πρώην σύζυγό του. Δεν έχει πολύ σημασία. Αυτό που βλέπουμε όμως να ισχύει είναι ότι πραγματικά ανώνυμες εταιρείε χρησιμοποιήθηκαν ως κρυψώνες και για παράνομα και για νόμιμα. Ευχαριστώ. Για το Βέλγιο υπάρχουν και ιστορικοί λόγοι για να προσπαθεί κανείς να κρύψει τα χρήματά του. Μια σειρά από ιστορικούς λόγους. Άννα Γκόμες για τους Σοσιαλδημοκράτες. Παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Η Μοσάκ Φονσέκα υποτίθεται ότι είναι η πρώτη από αυτές τις μεγάλες εταιρείες που έχουν ε, ε, ενορχιστρώσει ε, όλη αυτή την ιστορία με τις τράπεζές μας και τις εταιρείες offshore. Με τράπεζες, δικηγόρους, με χρηματοοικονομικούς ομίλους. Εσείς, για τις άλλες μεγάλες εταιρείες, τι μπορείτε να μας πείτε. Και επίσης προσπαθήσατε να, να ξεκριβώσετε αν υπάρχει ένα μοτίβο για τις ε, φορολογικές απάτες που έγιναν στα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια ως ένα τελευταίο βήμα για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος που κατευθυνόταν σε φορολογικούς παραδείσους όπως αυτούς που αποκαλύψατε. Για τα χρήματα αυτά, περιουσιακά στοιχεία που ήταν αποτέλεσμα φοροδιαφυγής ή διαφθοράς ή οργανωμένο εγκλήματος. Υπάρχει ένα μοτίβο. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεπλύνει κανείς το βρωμικό χρήμα. Σκέφτομαι ε, στην χώρα μου. Είχαμε τρεις περιπτώσεις φορολογικής αμνηστία. Ε, το 2005, 2008 και 2013 στην Πορτογαλία Ε, ήταν ε, αναγκαστικό να αποκαλυφθούν στοιχεία λόγω της Τρόικας και της ε, φορολογικής μας προσαρμογής. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν εδώ. Ευχαριστώ και αυτή η δύσκολη ερώτηση για τους δημοσιογράφους. Είναι μια ερώτηση που κυρίως πρέπει να απευθυνθεί στην Κομισιόν για τα κράτη μελά. Παρακαλώ. Θέλει κανείς να απαντήσει. Ε, προσφέρεται κανείς εθελουσίως. Ο κύριος Στρότσικ. Να προσπαθήσω να αναφερθώ στις ε, φορολογικές αμνηστίες ε, στη Γερμανία. Υπήρξε ένας διακανονισμός ε, για το ότι αν κάποιος αυτοκαταγγελθεί για φοροδιαφυγή τότε δεν έχει ποινικέ επιπτώσεις. Όπως είδαμε από τα έγγραφα, αυτά αφορούν άλλους ατόμους. άλλα άτομα, συγγνώμη. Κατά τη γνώμη μου, όποιος θέλει να φτιάξει μια εταιρεία offshore και τον βοηθά ένας δικηγόρος, μία τράπεζα. Αυτός θέλει να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν έχω στοιχεία, δεν έχω δημόσια στοιχεία, δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι αφορά άτομα που είχαν έναν απλό λογαριασμό στην Ελβετία ή κάπου αλλού για να πάνε χρήματα τα οποία δεν ήθελαν να εμφανιστεί ότι πάνε σε αυτούς. Βεβαίω θα προσπαθήσουμε να αποκαλύψουμε και άλλα δικηγορικά γραφεία που κάνουν τέτοιε δουλειέ, αλλά δεν είναι καινούργια αυτά τα πράγματα βεβαίω. Ούτε αυτά που κάνουν είναι καινούργια ω διαδικασία. Αυτέ οι διαρροέ μα επιτρέπουν όχι μόνο να δούμε συγκεκριμένα πώ γίνονται αυτά, αλλά μα επιτρέπουν να δημιουργήσουμε και ένα ενδιαφέρον. Γιατί είναι δύσκολο βέβαια να εντοπίσουμε παρανομίες, αλλά μας δίνεται η δυνατότητα να γράψουμε άρθρα για τα θέματα αυτά. Δεν είναι εύκολο να κάνεις καλό άρθρο μόνο με κάποια στοιχεία για το πώς λειτουργεί ένα δικηγορικό γραφείο. Πρόεδρος, ευχαριστώ το δεύτερο τμήμα της ε, ε, ερώτησης. Θα πρέπει να το συζητήσουμε κατά τη δεύτερη φάση των εργασιών μας με τις ε, αντίστοιχες αρχές και μάλιστα με πολύ προστατικό τρόπο. Κωνσταντζε Λεγκρίπ από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα του ερευνητέ δημοσιογράφου που απήντησαν στην πρόκλησή μα και μα έκαναν αυτέ τι παρουσιάσει. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε και πραγματικά διαφωτιστικέ. Νομίζω τώρα είμαστε σε θέση να καταλάβουμε ποια είναι τα μεγάλα δίκτυα και κλώματα που δημιουργήθηκαν, το σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο, το business plan για να το πω αλλιώ, που επέτρεψε αυτή τη φοροδιαφυγή και φοραπάτη για τη λεύκανση παράνομων προσόδων, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Βλέπουμε το κλασικό σύστημα ανώνυμες εταιρείε, ε, εικονικοί διευθυντές, δικηγόροι με αδιαφάνεια και ανωνυμία. Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά πολλά ήδη υπόθηκαν και κατά τη διάρκεια τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ποια είναι τα κενά και οι λήψει τη, τα δύναμα σημεία. Το κάλυψαν επαρκώς οι προλαλήσοντες συνάδελφοι. Ήθελα λοιπόν να επανέλθω σε ένα άλλο θέμα. Τους πληροφοριοδότες καταγγέλλοντες. Και εδώ πολλά υπόθηκαν. Και εσείς πρόεδρε, συχνά επιμείνατε στο ρόλο τους ποιες συγκεκριμένες δράσεις πρέπει να αναλάβουμε. Ποιες θεωρείτε ότι είναι συγκεκριμένες δράσεις που θα μπορούσαμε να ε, προτείνουμε στην λήψη μέτρων για την προστασία των καταγγελόντων. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω το έχουμε εξετάσει το θέμα ενδελεχώς, αλλά μπορούμε πάντα να έχουμε και άλλες απαντήσεις. Κύριε Τσίρμαν. Παρακαλώ. Δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά. Θα έπρεπε η νομοθεσία να τροποποιηθεί ώστε να μην υπάρχει κολασμός των ε, καταγγελόντων και επίσης το θέμα της διαφάνειας συνδέεται με το θέμα των ε, καταγγελόντων. Το είδαμε αυτό με το θέμα των τελικών των πραγματικών κατόχων, όπου είναι απαραίτητη η καταγγελία για να αποκαλυφθούν. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρξει τροποποίηση τη νομοθεσία ώστε να μην κινδυνεύουν να καταλήξουν στη στενή αυτή οι άνθρωποι, ώστε συγχρόνω να υπάρχει και η δυνατότητα εξασφάλιση τη διαφάνεια και η σωστή εφαρμογή τη νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό σίγουρα θα είναι πιο δύσκολο σε αυτέ τι συνθήκε να γίνονται πράγματα όπω αυτά που αποκαλύφθηκαν στα Panama Papers. Ευχαριστώ πολύ. Υπήρξε και ένα CD το οποίο είχε με τους Δανούς ε, πελάτες τραπεζών που ήταν το αποτέλεσμα της δράσης των ε, καταγγελόντων. Έχετε να θέσετε ένα ερώτημα περαιτέρω, κυρία Τεγκρύπ. Όχι, τότε έχει εξαρτηθεί ο κατάλογος των ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες. Έχουμε ελάχιστα λεπτά τώρα στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους διερμηνείς να μας δώσουν το πολύ 10 λεπτά πρόσθετα γιατί έχω άλλους επτά οι οποίοι βρίσκονται στον κατάλογο Catch the Eye. Ένα λεπτό το καθένα, ο καθένας σας. Ένα λεπτό λοιπόν ο Μπεντ Λούκε, η Φάμπιο Ντιμάση. Κύριος Μποργέτσο, Ματ ε, Κάρθη και η κυρία Νίουν Χρούζεν. Όλοι αυτοί είναι στον κατάλογο μου. Και μπορούμε να κλείσουμε τον κατάλογο μετά από όλα αυτά. Παρακαλώ, Μπέντλου και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημά μου αφορά τον κύριο Τσίλμαν. Αν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε, είπατε ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της και στις, ε, στα δικηγορικά γραφεία, γιατί δεν έχουν την ίδια ρύθμιση όπως ε, οι τράπεζες και είναι σε κάποια φαιά περιοχή πολλές φορές οι, οι δικηγόροι. Μιλάτε για τους δικηγόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάτε περισσότερο για δικηγόρους στην Ελβετία ή σε άλλες ε, περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιες είναι οι ρυθμίσεις που έχετε στο μυαλό σας, οι οποίες έχουν νόημα και για τις τράπεζες και για τις νομικές εταιρείες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός που θα εξασφαλίσουν περισσότερο τη διαφάνεια αυτή που λέτε. Τι ακριβώς θα μπορούσε να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε νομοθετικό επίπεδο για τον έλεγχο για τις ε, δικηγορικές εταιρείε οι οποίε δεν υπόκειται σε επαρκή έλεγχο. Κύριο Τσίρμαν, εγώ θα δώσω ένα ερώτημα. Εγώ μιλούσα για την Ελβετία. Οι δικηγόροι στην Ελβετία έχουν ένα σύστημα αυτορύθμισης σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Υπάρχει μια μορφή λοιπόν η οποία γίνεται σε επίπεδο επαγγελματικό από τους επαγγελματικούς φορείς τους. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της εργασίας της Μοσάκ Φονσέκα που γίνεται στην Ελβετία και ιδιαίτερα στην ε, Γενέβη. Και επομένως αυτά γίνονται στην Ελβετία. Τώρα για τους ε, Γερμανούς ε, δικηγόρους πολύ καλά, ξέρουν πολύ καλά οι συνάδελφοι από τη Γερμανία τι συμβαίνει και πώς ελέγχονται από την Μπάφιν. Μια σύντομη απάντηση η δική μου εμπειρία για τη Γερμανία δεν μπορούμε να συγχαίουμε το ρόλο των δικηγόρων με το ρόλο των τραπεζών. Ο Φάβιο από την ΚΟΕ. Ένα ερώτημα για τους συναδέλφους από το Αμβούργο. Έχετε φέρει πολλά άπλυτα στη φόρα. Και εγώ έχω ήδη προσπαθήσει να μάθω περισσότερα για τη Μόσακ Φονσέκα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στα νομοθετικά θέματα. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει μια νέα πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης είναι δυνατόν η, η εικονική ε, διευθυντές να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο όταν έχουμε ανοιχτά μητρώα για τους δικαιούχους. Και επίσης θα θέλατε να προβλεφθεί ένας ε, μαύρο, μια μαύρη λίστα για τις ε, χώρες όπου υπάρχουν ε, κάποιες ε, υπάρχουν εξωχωρές εταιρείε, αλλά αυτό θα πρέπει να περιβάλλει, να περιλάβει ίσως πολιτείες των ΗΠΑ όπως είναι η Νεβάδα και τον Τέλαγουα. Ποια είναι η αποψή σας λοιπόν για ένα πλήρη κατάλογο φορολογικών παραδείσων, κυρία Στάιν. Λοιπόν, πολύ σύντομα όχι στην πρώτη, ναι στη δεύτερη, όχι στην τρίτη ερώτηση. Άψογα κυρία Στάνιλη ο Πρόεδρος. Θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτό που μας είπατε για την περαιτέρω εργασία μας. Μόλις Σκοτ Κάρο Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ω ε, Βρετανή πρόσωπο. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο για αυτά τα θέματα τη φοροδιαφυγή. Ε, Κυρίω γιατί και η Βρετανία μπορεί να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνει μεγαλύτερο φορολογικό παράδεισο από τον κόσμο. Η υπόθεση του Panama Papers ω ε, Βρετανή Ευρωβουλευτού μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι οι περισσότερε από τι περιορισμένε εταιρείε ήταν καταγεγραμμένε στι Βρετανικέ νήσε τη Παρθένου. Με είχαν πολύ στενέ σχέσει με το Ηνωμένο Βασίλειο και το City του Λονδίνου, που είχαν τα περισσότερα δεδομένα. Ένα άλλο παράδειγμα ήταν οι Μπαχάμε, όπω αποκαλύφθηκε την περασμένη Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω του δημοσιογράφου αν συμμερίζετε την, την εντύπωσή μου ότι η Βρετανία ήταν μέρο του όλου θέματο αυτού και αν υπήρξε ε, μεγάλη ανάμεξη τη Μεγάλη Βρετανία ε, στην ε, ευρωπαϊκό σύστημα φοροδιαφυγή ή απλώς όλα παίρναγαν από την εταιρεία Mosaic Fonseca. Επίσης, ως προς την διαφάνεια, ε, η υπόθεση Panama Papers μας, εντόπισε, μας βοήθησε να εντοπίσουμε τους βασικούς παράγοντες και υπευθύνους εδώ. Τι πρέπει να γίνει για να νομοθετήσουμε και να δούμε την ακριβή θέση των Βρετανικών αρμόδιων φορέων. Σε Ενδιαφέρον το, το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου υπάρχουν και εκεί πολλές εταιρείες ε, γραμματοκιβωτίου. Ποιος θέλει να απαντήσει. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εταιριών που ήταν ε, καταχωρισμένες στις Βρετανικές Μητές Παρθένου. Όντως, ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι. Είναι εύστοχη λοιπόν η ερώτηση, διότι προηγουμένω κάποιο μίλησε για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Υπάρχει κίνδυνο τα κέρδη από τη φοροδιαφυγή να ε, προωθούνται μέσω του City του Λονδίνου, κάτι που έχουμε δει συχνά να συμβαίνει. Θα πρέπει εδώ να αναλυφθεί δράση από τους Βρετανούς, ώστε τα εξαρτώμενα εδάφη τους να λειτουργούν και αυτά με διαφάνεια. Είναι κέρια σημασία για τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστούμε, είσαι παπίτη Κάινον. Ευχαριστώ απλώς να υπογραμμίσω τη σημασία της προστασίας των καταγγελόντων και Ελπίζω σύντομα να βρούμε και να προτείνουμε κάποιο κανόνα. Πρέπει να έχει κανείς πληροφορίες ε, όταν ε, χρειάζεται να προστατεύσει συγκεκριμένε πρακτικές που είναι νόμιμες. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες από ό,τι κάνατε ως τώρα για την κλίμακα και δυνατόν για τη διασύνδεση των υποθέσεων μεταξύ τους. Με μια ιδιαίτερη μέρημνα στο που παρακάπτονται οι ευρωπαϊκοί νόμοι και κανόνες και που καταπατώνται τελείως. Και τρίτη ερώτηση, μπορείτε να δείτε κάποια διασύνδεση με τους πολιτικούς και την πολιτική υπονόμευσαν οι ίδιοι την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων κατά του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Και τελευταία μου παρατήρηση θα ήταν προβλέπεται ο να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για τα BEPS και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών εξαρκούν για να επιληθεί το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ποιος θα απαντήσει. Ορισμένα ερωτήματα έχουν βέβαια ήδη τεθεί. Κυρία Χνούς. Όχι. Well, the Η πρώτη ερώτηση είναι να μπορούμε, να μπορούμε σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Αυτή ήταν... Εάν μπορούμε να σας δώσουμε τα δεδομένα αυτό, είπατε. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να δώσετε όλες τις λεπτομέρειες. Απλώς ερωτώ εάν τα έχετε στα χέρια σας τα δεδομένα. Προφανώς δεν έχετε δημοσιεύσει τα πάντα ό,τι έχετε στα χέρια σας. Μπορείτε να μας δώσετε λοιπόν μια ανάλυση για να τα δούμε ως πολιτική, να δούμε που υπήρξαν παραβιάσεις της νομοθεσίας συγκεκριμένα έστω. Δηλαδή, αν μπορείτε να μα πείτε λίγο περισσότερο τι έχετε στα χέρια σα. Η απάντηση είναι ότι η ομάδα των αρνητών δημοσιογράφων έχει ήδη στον ιστότοπό τη ε, δημοσιεύσει ένα πολύ μεγάλο μέρο τη βάση δεδομένων μα, δεδομένα που έρχονται από τι διαρροέ του Panama Papers. Η απόφαση ήταν να μην μοιραστούμε τα 10.500 έγγραφα με τον υπόλοιπο κόσμο ε, κυβερνήσεις, φορολογικές αρχές κτλ. για τον απλό λόγο ότι είμαστε δημοσιογράφοι και ο ρόλος μας είναι να καταγγέλουμε ε, προς όφελος του κοινού, όχι να γίνουμε ε, καταγγέλλοντε και καταδότε κατά τη κυβέρνηση και τα διάφορα κοινοβούλια μας ζήτησαν να μην το κάνουμε, οπότε δεν ακολουθήσαμε αυτή την ακτική Τώρα για το αν οι ευρωπαϊκοί νόμοι παραβιάστηκαν ή καταπατήθηκαν ε, και πάλι, να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένω. Εάν υπήρξαν παραβιάσει, παρανομίε, νομίζω θα πρέπει να το δουν οι δικτικέ αρχέ και οι εισαγγελεί. Αυτοί να αναλάβουν δράση και να διώξουν. Κάποιε φορέ είναι πολύ λεπτό το όριο ε, και υπάρχουν γκρίζε ζώνε μεταξύ φοροδιαφυγή και φοροαπάτη. Η μία είναι νόμιμη, η άλλη είναι... μπορεί να είναι παρά, απλώς παράτυπη εφόσον είναι φοροαποφυγή. Πάντως, σε πολλά από τα άρθρα μας, ε, ε τα οποία προσκαλώ όλους να διαβάσουν στη γλώσσα τους και υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις. Μιλήσαμε με πυρογνώμονες παγκοσμίω για τα ζητήματα αυτά, οπότε ίσως ε, το καλύτερο είναι, σας παρακαλώ ευγενικά, να διαβάσετε όλα τα άρθρα που έχουν ήδη δημοσιευτεί. Ευχαριστώ. Σύρπα. Όχι, όχι, όχι, δεν έχεις άλλο χρόνο. Επόμενος. Να απαντήσω πολύ σύντομα. Είπατε ότι θέλετε περισσότερα έγγραφα. Στην πράξη, η δίκη που έχουμε στην Φιλανδία αυτή τη στιγμή έχει πολιτική πίεση από το Υπουργείο Οικονομικών, από το δικό σας κόμμα στη Φιλανδία. Ο Υπουργό σας το ξεκίνησε όλο αυτό και μας πήγε στα δικαστήρια. Οπότε οι φορολογικέ αρχέ μα το είπαν ανοιχτά. Έχουν πολιτική πίεση. Οπότε να το ξέρετε. Ευχαριστώ για αυτή την ε, σύσταση κύριε Ακνούς. Λοιπόν, τρεις ομιλίες. Ο κύριος Μποριέτσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μεταξύ των ονομάτων που δημοσιεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα ε, ε αναφέρεται και ο Τζοζέπε Ντονάλντο Νικοζία, ο οποίο είναι ένα από του μεγαλύτερου νονού τη Ιταλική μαφία, ο οποίο καταζητείται εδώ και χρόνια. Αυτό ε, είναι ένα σημαντικό μέρο τη έρευνά σα και θα ήταν ένα σημαντικό βήμα για να δοθεί συνέχεια στην υπόθεση Φαλκόνα Μπορσελίνο. Και βεβαίως ε, εδώ θα πρέπει ως ε, αρχή κατά πολέμηση του ξεκλήματος βρώμικου χρήματος να μην ε, παραμελήσουμε αυτό που μου είπαν και εμένα, ότι από τα ναρκωτικά τα βασικά κέρδη περνάνε μέσα από αυτό το δίκτυο που κατέληξε να είναι και το Panama Papers. Πώς λοιπόν θα διασταυρώσετε τα δικά σας δεδομένα για να τα αξιοποιήσετε σε συνεργασία με την άλλη αρχή στην Ιταλία που καταπολεμά το κύκλωμα της μαφίας. Ε, θέλει κανείς να απαντήσει, είναι κανείς σε θέση να απαντήσει, παρακαλώ κύριε Ζήλμαν. Δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορώ να μιλήσω για τους συναδέλφους στην Ιταλία, αλλά όπως και εμείς ψάχνουν για ονόματα συστηματικά και βεβαίως ε, δεν μας εκπλήσει το ότι υπάρχουν και εκπρόσωποι και ηγέτες και καταδικασμένοι του οργανωμένου εγκλήματος. Αλλά βέβαια δεν έχουμε πλήρως ε, εξετάσει αυτό το υλικό ε, είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολλές σελίδες. Κάθε φορά που ξαναμπαίνει κανείς να διαβάζει βρίσκει και άλλα ονόματα και άλλες λεπτομέρειες. Ε, διαπιστώνεις για παράδειγμα ότι δεν έχουμε βρει όλα τα άτομα που έχουν παίξει αποφασιστικό ρόλο. Άρα νομίζω ότι έχουν κάνει πολλά οι συνάδελφοι στην Ιταλία. Μακάρθι. Από την ΚΟΕ ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εύχομαι στην κυρία Κνούς και, την, και στο φορέα της κάθε επιτυχία στον αγώνα για να διατηρήσουμε τις ελευθερίες μας. Αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει είναι πόσες φορολογικές αρχές σε όλη την Ευρώπη δεν έχουν καταβάλει καμία απολύτως προσπάθεια για να φτάσουν στην πηγή του κακού και να αποκτήσουμε πληροφορίε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εταιρείε όπω η Mossack Fonseca χρησιμοποιούνται από δικτάτορε, από μαφίε. Οι περισσότεροι άνθρωποι όμω που χρησιμοποιούν αυτή την εταιρεία είναι αυτοί που θεωρούσαμε ότι είναι οι κολόνες της κοινωνίας μας και παρόλα αυτά εμπλέκονται σε αυτή την συστηματική κλοπή πλούτου της κοινωνίας μας με φοροαπηφυγή και φορο διαφυγή. Το ερώτημα που θέλω να θέσω λοιπόν σε δημοσιογράφου είναι πώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που έχετε εσείς για να μπορέσουμε να δώσουμε στοιχεία στι φορολογικέ αρχέ συγχρόνω προστατεύοντα την ελευθερία των δημοσιογράφων και να κάνουμε αυτό που φοβούνται περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι μονάχα να τους αποκαλύπτουμε, αλλά το να του υποχρεώσουμε να πληρώσουμε το φόρο που οφείλουν στις φορολογικέ μα αρχέ. Ευχαριστώ. Ήταν περισσότερο μια δήλωση. Κυρία Κνούτ, θέλετε να πείτε κάτι. Όπως είπαμε και προηγουμένως, όλα αυτά που δημοσιεύουμε είναι πραγματικά ενδιαφέροντα για τις φορολογικές αρχές να τα εξετάσουν όλα αυτά τα στοιχεία για τις εταιρείε offshore αλλά είναι διαθέσιμα. Ξέρω ότι ο ανώνυμος αυτός καταγγέλων είπε ότι ήταν έτοιμος να συνεργαστεί με τις φορολογικές αρχές. Δεν ξέρω αν υπήρχε σε κάποια αίτηση προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά και αυτό θα ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, πιστεύω. Ευχαριστώ. Τελευταία. Η κόρα να από την άλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες εδώ και συζήτησαν μαζί μας τόνισαν όλοι οι δημοσιογράφοι την ανάγκη να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή του νόμου. Θέλω να θέσω το εξή ερώτημα. Υπήρχε μια υποχρέωση για τι τράπεζε να αναφέρουν όλες τις ύποπτες δοσοληψίε. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ελέγξουν και αναδρομικά τι υπήρξε. Υπήρξαν όμως περιπτώσεις όπου είχατε στοιχεία ότι τέτοιου είδου ύποπτες συναλλαγέ δεν ε, αναφέρθηκαν και αντίθετα υπήρξε κάποια εμπλοκή τραπεζών σε διαφθορά ή σε έκπληση χρημάτων. Ποιος θα ήθελε να δώσει τις τελευταίες απαντήσεις. Κύριε Κλούς, ναι. Η απάντηση είναι ναι. Ναι, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις, ιδίως άμα δείτε τις εκθέσεις από τα Βρετανικά νησιά της Παρθένου. Υπήρξαν ακόμα και περιπτώσεις όπου αναφέρθηκαν ύποπτες συναλλαγές, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια έχουν πουληθεί εταιρείε offshore σε ένα καταδικασμένο παιδόφιλο ο οποίο είχε οργανώσει ένα δίκτυο παιδοφίλων και αυτό δεν, είχε, δεν έτυχε καμία συνέχεια, δεν υπήρξε δίωξη η οποία έγινε στη συνέχεια, δεν έγινε καμία προσπάθεια εφαρμογής αρχής τη πρέπει σας επιμέλειας. Αυτό ίσω είναι μια απάντηση στο ερώτημα τη κυρία Κνιχάιζεν. χωρί ε, ο μικρόφωνο πρόεδρο. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτήν την συνεδρίαση και συνεργάστηκαν μαζί μας και τους δημοσιογράφους δυστυχώς δεν καταφέραμε να συνεννοηθούμε με τον κύριο Όμπερ Μάιρ Ελπίζω ότι θα έχουμε και κάποια ευκαιρία στο μέλλον να τον ακούσουμε ως ένα από τους ε, ε δημοσιογράφους που απεκάλυψαν όλα αυτά τα στοιχεία. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους συναδέλφους. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά και σημαντικά και ακούσαμε τις προτάσεις για πολλά μέτρα τα οποία πρέπει να αναλυθούν. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα λοιπόν και αυτή η ακρόαση θα είναι πολύ χρήσιμη για να έχουμε και περαιτέρω επεξεργασία των θεμάτων Θέλω να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς και τη γραμματεία για την προετοιμασία αυτής της συνεδρίασης και να σας προσθέσω ότι η Προεδρία, το Προεδρείο μας μαζί με τους δύο εισηγητές θα είναι διαθέσιμο για τους δημοσιογράφους αν θέλουν να μας θέσουν ερωτήματα. Κλείνω τη συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα για όλους.